Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Εάν μου δώσει την ευκαιρία ο κύριος Γκάλα. Ευχαριστώ. καλωσορίσω τον πρόεδρο της Επιτροπής για το Ανθρώπινα Δικαιώματα του Βιετνάμ. Δράση για τη δημοκρατία στο Βιετνάμ, τον κύριο Φο Βαν Χάι. Θα συνοδεύει η κυρία Φόκνερ. Καλώς ήρθατε. και ο κύριο Ζωμαρί Γουζ εκπροσωπεί τη Διεθνή Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την οργάνωση για την ελευθερία του διαδικτύου και την απελευθέρωση των blogger που βρίσκονται στη φυλακή στο Βιετνάμ. Καλώ ήρθατε και ελπίζω να σας ενδιαφέρουν οι εργασίες μας. Κυρία Φούκνερ. Θα έχει την ευκαιρία κάποιων επαφών μαζί μας. και θα μας ενημερώσει για τα θέματά της. Παρακαλώ να αφήσετε ανοιχτές τις πόρτες για να την υποδεχθείτε. Στο σημείο 3. Πρακτικά τη συνεδρία αυτή και 7η συνεδρία. Όσοι τα έχουν διαβάσει μπορούν να τα εγκρίνουν. Οι λοιποί μπορούν να τα καταψηφίσουν. Δεν βλέπω να κινείται κανεί, άρα εγκρίνονται. Και τώρα Περνάμε στο θέμα της Βόρειας Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο κύριος Φαρέλ θα μας ενημερώσει. γιατί φαίνεται ότι η Βόρεια Κορέα, όπως καταγράφεται, ε, α, εξακολουθεί να απειλεί την ασφάλεια των γειτόνων της, α, εξαπολύει απειλές ότι θα εξολοθρεύσει τη Νότια Κορέα και γίνεται έκκληση για μια διεθνή συνέλευση. Είχαμε μία δοκιμή από πλευρά τη Βόρεια κορέα από δύο εβδομάδε. έχει καταδικαστεί απερίφραστα από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά εξακολουθεί η Βόρεια Κορέα να ισχυρίζεται ότι είναι σε θέση να θέσει, να εκτοξεύσει πύραυλο με πυρηνικά και σκεφαλές. Ενδέχεται η κινητικότητα που εμφανίζεται να δείχνει τάσεις για ε, εντατικοποίηση των πυρηνικών εξοπλισμών. Περιμένουμε βέβαια να δούμε και τις εξελίξεις με την ανάληψη της εξουσίας από τον νέο γιατί Κιμ τις την αντίδραση της Κίνας και τις περαιτέρω εξελίξεις. Περιμένω να ακούσουμε τα θέματα αυτά λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον γιατί μπορεί αυτή η κατάσταση να έχει περαιτέρω εξελίξεις. Κύριε Στάνοκ, κύριε Πρόεδρε, περίμενα ότι θα ανακοινώνατε μεταξύ άλλων ότι ένας από τους ε, Ξέρετε, ο συναδέλφους, διορίστηκε υπουργό των Εξωτερικών, ο κύριο Κασουλίδη στην Κύπρο. Περιμένω ότι θα το ανακοινώνατε και ότι θα τον, συνεχέρε, θα τον συγχαρόσασταν για, τις, ε, για την ανάπτυξη των καθηκόντων του. Ναι, κοιτάξτε κύριε Τάνακλη, ο προεδρό. Ε, εγώ αποφασίζω ότι θα πράξω. Σα ευχαριστώ που διαβάσατε τι εφημερίδε. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φαμπρίς Φαρέλ. Um, uh, Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να ενημερώσω την Επιτροπή σας για τις τελευταίες εξελίξεις ε, στην Βόρεια Κορέα και για τις, ε, την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δώσατε μια καλή περιγραφή της κατάστασης έχει δημιουργήσει διαδοχικούς κύκλους αντιπαράθεσης με κύκλους ύφεση και καταλλαγής η Λαϊκή Κορέα, η Βόρεια Κορέα, ανάλογα και με τις ε, αλλαγές της εξουσίας στις γειτονικέ χώρες. Ξέρετε ότι έχουν υπάρξει πάρα πολλές αλλαγές ε, στη Νότια Κορέα, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, <clears throat> πολιτικές αλλαγές και αυτό το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας για να δυσκολεύει εξ αρχής τις ε, νέες κυβερνήσεις αυτών των χωρών. Αυτό που, συνδέεται, που γίνεται τώρα λοιπόν στην Βόρεια Κορέα εξαρτάται ίσως από αυτό το οποίο είπα. Υπήρξε μια ελπίδα ότι ο Κιμ Ιου Χουν, ο οποίος διεδέχθη τον πατέρα του πριν ένα περίπου έτος, θα οδηγούσε σε κάποιες θετικές αλλαγές στη χώρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δυστυχώς όλα αυτά πλέον εξανεμίστηκαν. Κανείς δεν συζητάει για οικονομικές μεταρρυθμίσεις και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ε, επιστροφή σε μια αποκλειστική εξάρτηση από τη στρατιωτική εξουσία. Ε, ξέρετε ότι η εκτόξευση του λεγόμενου αυτού ε, δορυφόρου δεν ήταν παρά ένα τεστ βαλιστικής τεχνολογίας. Ακολουθήθηκε από αυτή την πυρηνική δοκιμή πριν δύο εβδομάδες παρά τις τεράστιες εκκλήσεις ε, της διεθνούς κοινότητας να μην προχωρήσει σε αυτή τη δοκιμή. Δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες της συγκεκριμένης δοκιμής. Όπως είπατε, το μέγεθος ανταποκρίνεται σε ένα σεισμικό συμβάν. Αυτό σημαίνει ότι η έκπληξη ήταν ισχυρότερη από τις δύο προηγούμενες, το 9 και το 6. Οι δύο προηγούμενες δοκιμές πιστεύετε ότι χρησιμοποίησαν καύσιμο πλουτονίου. Ξέρετε ότι το 2010 ήρθε στην επικαιρότητα το ότι η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιούσε, προωθούσε πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου και αυτό οδήγησε στην προβληματική αν θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τέτοιου είδους όπλο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε ίχνη για το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην πρόσφατη δοκιμή. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογήσει κανείς είναι η ικανότητα της Βόρειας Κορέας να σχεδιάσει ε, ε, ε, ένα μηχανισμό αρκετά ελαφρύ που να μεταφέρεται με βαλιστικό φορέα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε, ξέρουμε πράγματι ότι πρόκειται για στρατιωτικής υφής και χρήσης υλικό αυτό που χρησιμοποιήθηκε, αλλά δεν ξέρουμε τα τεχνικά όρια της Βόρειας Κορέας. Αυτό είναι μια περαιτέρω παραβίαση των διεθνών ανηλυμένων υποχρεώσεων της Βόρειας Κορέας σε σχέση με το σεβασμό των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει τους κινδύνους που παρουσιάζει το πρόγραμμα αυτό πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας και αυξάνει την ικανότητα ε, της Βόρειας Κορέας να στρατιωτικοποιήσει τους πυρηνικούς μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή της. Αυτό δημιουργεί περαιτέρω εντάσει στον Νοτιοανατολική Ασία και αυτό είναι ένας επιπλέον παράγωνα ε, περιφερειακής αστάθειας. Κάτι το θετικό που μπορεί κανείς να υπογραμμίσει ήταν η ενωμένη ανταπόκριση της διεθνούς κοινότητας στην αντίδρασή της. Άνω των 80 χωρών εξέδωσαν δηλώσεις ανακοινοθέντα που καταδικάζουν την δοκιμή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι η διεθνής κοινότητα συνεχίζει ενωμένη να καταδικάζει τις ενέργειες της Βόρειας Κορέας. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκάθαρα και με ταχύτητα καταδίκασε όλες τις τελευταίες, τις πρόσφατες καταδικαστές ενέργειες της Βόρειας Κορέας. Η κυρία Άστον και πριν και μετά από την εκτόξευση του δορυφόρου εξέδωσε ανακοινοθέν. Εξεδόθη επίσης και ένα ανακοινοθέν από πλευράς ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και μετά από την πυρηνική και πριν και μετά από την πυρηνική δοκιμή και αυτό συνοδεύθηκε με ένα κείμενο καταδίκης α, ε, της 18ης Φεβρουαρίου. Έχει μεγάλη σημασία να υπογραμμίσουμε εδώ ότι το βασικό ε, πρόβλημα ε, μιας ε, ελεύθερης από πυρηνικά Χευσονήσου είναι η Βόρεια Κορέα. Ε, δεν αρκεί οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία να καταδικάζουν βέβαια τη δοκιμή, αλλά έχει ενδιαφέρον να βλέπει κανείς ότι υπήρξε μία χωρίς καμία διαφοροποίηση καταδίκη από πλευράς της λαϊκής Κίνας, παράλληλα με την καταδίκη της διεθνούς κοινότητας. Συνεπώς η κινέζικη καταδίκηση συνιστά μια αλλαγή τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσίου μηνύματος αν θέλετε γύρω από το ποια είναι η θέση της λαϊκής δημοκρατίας. Δεν είναι ξεκάθαρο βέβαια εάν αυτό ε, θα οδηγήσει σε μια αλλαγή πολιτικής ε, την οποία θα ασκεί η νέα κυβέρνηση στο Πεκίνο. Τώρα, οι βασικοί πρωταγωνιστές βέβαια στην καταδίκη ήταν τα Ηνωμένα Έθνη και οι Ηνωμένε Πολιτείες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είπε ότι θα προχωρήσει, θα προτείνει νέα μέτρα στα πλαίσια των συζητήσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά από την εκτόξευση του δορυφόρου χρειάστηκε ένας μήνας για να καταλήξουμε σε μια συνένεση και με την Κίνα και σε αυτή την περίπτωση επίσης θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έτσι ώστε να καταλήξει το Συμβούλιο Ασφαλείας σε ένα ουσιαστικό μήνυμα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καταρχάς ε, είναι υπέρ ε, μιας μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας το σύστημα διεθνών κυρώσεων επί τη βάση συγκεκριμένων νομικών διεθνών συμβάσεων. Το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα πρώτο πακέτο μέτρων στις 18 Φεβρουαρίου εφαρμόζοντας τις προβλέπεις οι οποίες προβλέπονται από το προηγούμενο ψήφισμα του μηνός Ιανουαρίου του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπάρχουν και κάποια επιπλέον δεσμευτικά περιοριστικά μέτρα σε σχέση με τον οικονομικό τομέα ή σε σχέση με την εξαγωγή κάποιων βασικών υλικών για την κατασκευή τέτοιου είδους βλημάτων βασική αλλαγή θα έλεγα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η συνεργασία με χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα αυτή τη φορά που και οι δύο αυτές χώρες παίζουν ένα κομβικό ρόλο στα πλαίσια της προετοιμασίας και της εφαρμογής μιας αξιόπιστης και αποτελεσματικής διεθνούς ανταπόκρισης. Πέραν τούτου, εξακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί και την εξέλιξη στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην λαϊκή δημοκρατία της Κορέας. Ξέρετε ότι υπάρχουν βαρύτατες παραβιάσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει ένα ψήφισμα στο επίπεδο του Συμβουλίου Ασφαλείας έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Βόρεια Κορέα. Αυτά. Κύριε Gomes. ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Υπηρεσία Υπηρεσίας δράση Δράσης για την ενημέρωση αυτή. Θεωρώ ότι στην τελευταία σειρά σοβαρών αυτών ε, προβλημάτων και προκλήσεων από τη Βόρεια Κορέα. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά να περάσουν παρατηρήτα. Δεν επαρκεί να τα καταδικάζουμε αυτά σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις αυτές που έχουν γίνει. Αυτό επηρεάζει ασφαλώς τη δυνατότητα της ε, Βόρειας Κορέας ε, για τα πυρηνικά και για την ε, διάδοσή τους και για την ε, κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ε, Βόρεια Κορέα. Όλοι ξέρουμε ότι είναι απαράδεκτα τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι που θα εμποδίσει τις δράσεις της ηγεσία αυτής. ώστε να μην μπορέσει να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο η ηγεσία της Βορειοκορέας. Νομίζω ότι πολλοί εξημών, πολλοί εδώ στην Ευρώπη και ίσως και στη ΣΥΠΑ, ίσως να θεωρούσαν ότι η Κίνα θα μπορούσε να τα ε, κρατήσει υπό έλεγχο τα πράγματα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το καταφέρνει αυτό, γιατί η Κίνα σήμερα καταδικάζει στο ε, Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει οτιδήποτε, δεν μπορεί να σταματήσει το οτιδήποτε και ενδεχομένω να μην μπορέσει να αποτρέψει και τις μελλοντικέ εξελίξεις. Ερωτώ λοιπόν τον εκπρόσωπο της υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι το εξή, Ρωτώ το εξής. Πώς ε, αξιολογούμε το ρόλο της Κίνας, φυσικά η αντίδραση της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ, της Νοτιού Κορέας. Ήταν αυτές που ήταν οι αναμενόμενες δεν έχουν ασφαλώς και αντίκτυπο ιδιαίτερο στην ε, Βόρεια Κορέα. Η Κίνα είναι αυτή που έχει σημασία. Τι λέμε λοιπόν προς τους Κινέζους, τι περιμένουμε από αυτούς. Τι προπτικές υπάρχουν σε ό,τι αφορά την μελλοντική επιρροή της Κίνας για να συνεφέρει κάπως την ηγεσία της ε, Βορείου Κορέας και να την πείσει να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κατσίν. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό που γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψε. αλλά δυστυχώς Όσο τέτοιου είδους συζητήσεις είναι ανοιχτέ προς το κοινό, δεν μπορούμε να αναμένουμε να ακούσουμε κάτι σημαντικό ή ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε οποιαδήποτε συμφωνία για τα περαιτέρω Γιατί το θέμα δεν είναι ποιος είναι ο ρόλος της Κίνας. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός ε, των πυρηνικών αυτών δοκιμών. Και αυτό μπορεί να συζητηθεί μόνο αν έχουμε στη διάθεσή μας και τα σχετικά στοιχεία. Ο νέος ηγέτης είναι καινούριο. Μπορούμε να κάνουμε διάφορες εικασίες για το τι πραγματικά πράττει και τι κάνει. Κατά πόσον ε, ε, απειλεί οποιονδήποτε άλλο πέρα από τη Βόρεια Κορέα ή κατά πόσο προσπαθεί να ελέγξει πλήρως το στρατό, αν προετοιμάζει το κράτος για τις ε, μεταρρυθμίσεις που κατεπηγόντως χρειάζεται και προς τα ποια κατεύθυνση θα στραφούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ επίκαιρα, χωρίς όμως βαθύτερη ανάλυση και σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις. Μπορούμε να καταδικάζουμε μεν και να επιβάλλουμε κυρώσεις, οι οποίες όμως δεν ξέρουμε κατά πόσον θα είναι καρποφόρες, κατά πόσον θα πετύχουν αυτό που επιδιώκουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα κάτι παραπάνω. Θα ήθελα να ακούσω πιο πολλές λεπτομέρειες, πιο πολλά επιχειρήματα και καταρχάς στοιχεία, με λιγότερα αν, αν θέλετε, σε σχέση με αυτά που έχουμε, αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αν είναι τόσο αδύναμη, αν θέλετε, και σαφρή η ανάλυση μας, καλό ίσως θα ήταν να έλθουν εδώ ε, υπουργοί από τα κράτη-μέλη που έχουν ε, πρεσβείες στην Βόρεια Κορέα και μπορούν επιτόπου από πρώτο χέρι να μας πούν τι γίνεται. Δεν ε, παραπονιέμαι, απλά διαπιστώνω ότι αυτά που ακούσαμε δεν επαρκούν για οποιαδήποτε ανταλλαγή απόψεων. Πόσο μάλλον για οποιαδήποτε εξαγωγή συμπερασμάτων ή συστάσεων. Μιλάμε σε θεωρητικό επίπεδο. Δεν είναι ο ρόλος αυτός της Ευρωπαϊκής σε ό,τι αφορά τέτοια σημαντικά θέματα και τόσο σημαντικές προκλήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος um, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κατσίν, κοιτάξτε, αν ε, ήταν και κλεισμένο των θυρών η συνεδρίαση αυτή, δεν θα ακούγατε και τίποτα περισσότερο, γιατί οι συνεδριάσει και κλεισμένων των θυρών στο Κοινοβούλιο δεν λένε τίποτα περισσότερο από ό,τι λένε οι εφημερίδε. Εν πάση περιπτώσει, η τρίτη γενιά των Κιμ είναι εξίσου κακή με τον παππού του. Ε, καταδικάζω την Βόρεια Κορέα εδώ και δέκα χρόνια σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο και δεν έχει συμβεί εις βάρος της τίποτα. Είναι μια πρόκληση η πυρηνική αυτή δοκιμή Τώρα έχει ένα πρόγραμμα παράλληλο και με πλουτόνιο και με ουράνιο και προφανώς θα καταφέρουν ε, να προχωρήσουν στην στρατιωτική ε, χρήση της βαλιστικής τεχνολογίας, ίσως όμως όχι ακόμα με υπερπόντια δυνατότητα εμβέλειας. Ε, το καθεστώς των κυρώσεων για μια ακόμη φορά θα είναι ανεπαρκές αυτό που έγινε οφείλεται στην ενθρόνηση σε εισαγωγικά του νέου Προέδρου της Νότιας Κορέας και τέτοιες αντιδράσεις δεν είναι καθόλου ορθολογικές και είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό το οποίο συμβαίνει, μόνο και η λαϊκή Κίνα κάτι μπορεί να κάνει, αλλά όχι και πάρα πολλά, έτσι ώστε να οδηγήσει το καθεστώς της Πνόγγιανγκ στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Και ίσως μια ελπίδα να έγκυται και στο ότι δεν θα αντέχουν πια οι κάτοικοι της Βόρειας Κορέας την κατάσταση, αλλιώς φοβάμαι δεν θα αλλάξει τίποτα όπως δεν άλλαξε τα τελευταία δέκα χρόνια. Ευχαριστώ. Κύριε Κασίνη, έχετε δίκιο. Και σε κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίες δεν θα μαθαίναμε περισσότερα από ότι σε μια δημόσια, γιατί τους άλλους δεν ξέρουν τίποτε περισσότερο αυτοί που έρχονται να μας μιλήσουν. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου μόνο γενικέ εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Εκτός πια και αν αρχίσουμε βέβαια τις υποθέσεις ε, να διαβάζουμε τα άστρα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, ο καθένα έχει από λίγα στοιχεία. Αναφερθήκατε εσεί ήδη ότι μπορεί να υπάρχει δυνατότητα η Βόρεια Κορέα να εμφανιστεί με τη νέα της ηγεσία πολύ πιο ε, φανερά στο διεθνές προσκήνιο να προσπαθήσει να διεκδικήσει πιο ισχυρή θέση και ενδεχομένως να είναι και διατεθειμένη για περισσότερους συμβασμούς. Αλλά με τις ελπίδες αυτές Πολλές φορές έχουμε διαψευστεί από τέτοια καθεστώτα. Ίσως είναι και αυτό μια δυνατότητα ωστόσο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Όμως αποτελέσματα θα δούμε μόνο εάν οι δράσεις που διαπιστωμένα έχουν λάβει χώρα ε, συναντούν και την αντίστοιχη αντίδραση για να είναι κατάσταση. Γιατί πολλές φορές έχουμε κάνει υποθέσεις ε, ή προβλέψεις ή εκτιμήσεις ε, οι οποίες έχουν ε, διαψευστεί ξαφνικά με την εμφάνιση είτε μιας βόμβας είτε πυράβλων. Δεν νομίζω ότι έχουμε περιθώριο να κάνουμε τέτοια σφάλματα πλέον. και να βρεθούμε ενώπιον μιας, ε, ε, της παραγωγής μιας βόμβας σε ενός πυράβλου μεγάλου Εάν δεν δούμε στην ευρύτερη περιοχή την κρίση μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας, εάν δούμε την κατάσταση μεταξύ Ινδονησίας και Φιλιππινών, εάν όλα αυτά και ε, εντάξουμε στην εικόνα και το Ιράν με την ε, χειρότερη δυνατή εκδοχή να εξοπλιστεί και το Ιράν με πυρηνική βόμβα, τότε βλέπουμε ότι όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ εκρηκτικό, ε, ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα. Και βέβαια αυτό ε, ίσως να εμπνεύσει και άλλες περιφερειακές δυνάμεις να εξοπλιστούν με πυρηνική βόμβα. Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, για να αναφερθώ και στη Μέση Ανατολή ε, που θα μπορούσαν ενδεχομένω να εμπνευστούν. Και έτσι, σε αυτό το χειρότερο δυνατό σενάριο, αποτυγχάνει η, ε, το σύμφωνο μη διαδόσεως των πυρηνικών και ο εξοπλισμός με πυρηνικό όπλο καθίσταται κάτω τετριμένο και κοινό. Για οποιονδήποτε μπορεί να εξασφαλίσει βέβαια ε, τα όπλα αυτά. Ε, με αυτή την έννοια λοιπόν έχει πολύ δραματικό χαρακτήρα αυτή η εξέλιξη στην Βόρεια Κορέα και κυρίως δεδομένων των εξελίξεων στην περιοχή αυτή. Όπως είπα, εάν ε, το συνδυάσουμε με την ε, μεγάλη ε, κλιμάκωση στους ναυτικούς εξοπλισμούς αλλά και στο στρατό στην Κίνα ενδέχεται πολύ γρήγορα να διαπιστώσουμε μια ριζική ανατροπή της κατάστασης στην περιοχή. Δεν είμαι δε ότι έχουμε ε, προετοιμαστεί και ότι ε, οι συνθήκες είναι αντίστοιχε με αυτές που είχαμε πριν από 60 χρόνια και την ε, διέρεση του κόσμου σε μπλοκ. Είναι τελείως διαφορετικές ισορροπίες δυνάμεων τώρα και οικονομικές, όχι μόνο στρατιωτικές. Μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ ριζικές ανατροπές και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θέλει κάποιος άλλος ε, από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να πει κάτι ακόμη. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Αναφερθήκατε την γιαγκολογία ε, ή διατηνομολογία είναι δύσκολη αυτή η επιστήμη, δύσκολο να συλλέξει κανείς στοιχεία στη Δύση. Οτιδήποτε πούμε είναι απλώς υποθέσεις. Έχουμε κάποια κρατημέλη με εκπροσώπηση στην Πιονγκιάνγκ που μας ενημερώνουν μέσα των αντιπροσωπιών τους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των σχέσεων. Δεν συμμετέχουμε στις εξαμερείς συνομιλίες, δεν έχουμε παρουσία με δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή αυτή του κόσμου ε, και ως εκ τούτου προσπαθούμε απλώς να συμβάλλουμε όπως πάντα στην αποτροπή των ε, κλιμακώσεων και των βαλιστικών πυράβλων, ε, δηλαδή την αποτροπή των μέτρων που στόχο έχουν την ενίσχυση των εξοπλισμών. Για δε την Κίνα, όπως και εσείς ε, αλλά και άλλοι συνάδελφοι σωστά επισημάνατε, έχει κρίσιμο ρόλο εδώ να διαδραματίσει η Κίνα. Αναφέρεται ότι έχει ασκήσει πολύ σημαντικές πιέσεις στη Βόρεια Κορέα η Κίνα να μην διαξαχθούν τον Φεβρουάριο οι προγραμματισμένες δοκιμές, ωστόσο η ε, Βόρεια, η Βόρεια Κορέα δεν ε, υπάκουσε και προχώρησε στις δοκιμές της, ως εκ τούτου φαίνεται ότι είναι περιορισμένη η επιρροή που μπορεί να έχει η Κίνα στη Βόρειο Κίνα, με συνέπεια εν τέλει μια μετριοπαθή καταδίκη από πλευρά της Κίνας, της Βόρειας ε, Κορέας για τις δοκιμές αυτές. Μια καταδίκη η οποία ίσως δείχνει μια με καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν απόσταση της Κίνας σχέση με τη Βόρεια Κορέα. Αλλά πάντως εμείς ε, αυτό που ε, μας κάνει να συγχωρούμε ιδιαίτερα είναι ότι ένα καθεστώς με αντιδράσεις τόσο απρόβλεπτες όσο αυτές της Pyongyang ενδέχεται να εξοπλιστεί με ε, Τέτοια αποτελεσματικότητα όπλα, το ίδιο βέβαια ανησυχεί και την Κίνα, είναι πιθανόν ε, να βρίσκονται και εκείνοι σε πολύ δύσκολη θέση γιατί δεν έχουν στα χέρια του καλά χαρτιά, δεν έχουν λύσεις ε, αίσιες. Κάποιος από τους βουλευτές αναφέρθηκε στην κυρία Πάρκ και τα σημερινά εγγένεια που έγινε λόγος για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου. Και περιμένουμε να δούμε αυτές οι προσπάθειες, αυτή η νέα πολιτική ε, της Σεούλ, τι είδους αντιδράσεις θα φέρει από πλευράς της Βόρειας Κορέας. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Κατσίν, ευχαριστώ πολύ. Ναι, να απαντήσω σε αυτά που δήλωσε η Επιτροπή. Ως τώρα όλες οι προκλήσεις, οι πρινικές δοκιμές και τα λοιπά χρησιμοποιήθηκαν για τον ένα και αυτό σκοπό. Για να ανανεώσουν το διάλογο με την Βόρειο Κορέα. Και ένα από αυτά τα σχετικά φόρα είναι η εξαμελής συζητήσεις, αυτές τις συζητήσεις των έξι ημερών, πάντα ζητούν να καταστούν σημαντικοί φορείς. Το θέμα όμως είναι πώς θα αντιδράσουμε εμείς. Θα διαδραματίσουμε ρόλο στις ε, ενδεχόμενε μελλοντικέ ε, συζητήσεις στα πλαίσια της εξαμερούς αυτής της ομάδας ή θέλουμε να είμαστε παρατηρητές από, τα από μακριά όπως τώρα θα ήθελα να πω ότι αυτή η συζήτηση, αυτή η ανταλλαγή απόψεων εδώ στο Κοινοβούλιο νομίζω ότι καταδεικνύει τις ικανότητές μας. Και η εικόνα που, συνθή, δεν είναι πολλά υποσχόμενη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταστούμε πολύ σχετικώς ε, παράγοντας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία απάντηση. Θα απαντήσουμε θετικά σε περίπτωση που θέλουν να συμμετάσχουμε στο διάλογο ή όχι. Κύριε Κασίν, ξέρω ότι έχετε τις καλύτερες των προθέσεων. Εγώ παρακολουθώ τα θέματα της Λαϊκής Κορέας εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Η Λαϊκή Κορέα δεν ξέρει ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ενδιαφέρεται για την Ευρώπη. Αν έχει κάποιο νόημα αυτό που κάνουν, που δεν έχει συχνά, είναι εις βάρος των Αμερικανών. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς αντιδρούν οι Αμερικανοί, τίποτα άλλο. Τώρα αν είμαστε ε, μέσα στις διαπραγματεύσεις της εξαμερής και τα λοιπά, δεν θέλω να σας απογοητεύσω κύριε Κασίνα, αλλά αυτό είναι ε, σαν να βαφκαλιζόμεθα. Η άλλη πλευρά δεν ενδιαφέρεται. Δεν έχουν καν αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Έχουν μία αντιπροσωπεία στην Ευρώπη και αυτή βρίσκεται στο Βερολίνο. Αυτό είναι το μοναδικό τους ενδιαφέρον για την Ευρώπη. Κύριε Τάνοκ, μιλήσατε... Μιλήσατε για πράγματα τα οποία υποστηρίζω, που ενδεχομένω να υποστηρίζουμε και δεν θα ήθελα να τα υποστηρίζω. Δεν νομίζω ότι είναι η παρούσα χρονική στιγμή να αλλάξουμε το μορφότυπο των διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι έχει ρόλο για την Βόρεια Κορέα και αυτό το γνωρίζω από πολλές επαφές στην, ε, με τη Βόρεια Κορέα. Και σκέφτομαι στην παρούσα φάση, ίσως θα μπορούσαμε να το κοιτάξουμε και σε πλαίσιο των ομάδων στην ε, Βόρεια Κορέα και σε ό,τι αφορά την φάση της ε, ανάπτυξης του Ιράν. Η κυρία Άστον θα είναι το Μάρτιο στο Στρασβούργο και τώρα έχουμε το θέμα της μη διάδοσης. Είναι μήπως θέμα για να το θέσουμε στο Στρασβούργο. Μήπως οι ομάδες θα ήθελαν να το συζητήσουν αυτό στο ιστορικό τους και ίσως θα μπορούσαμε εκεί να κάνουμε την ενδιαφέρουσα αυτή τη συζήτηση και να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις, τις σημαντικές αυτές εξελίξεις. Δεν ξέρω τι λέτε. Αν το θέλετε, συζητήστε το με τους συντονιστές και θα μπορέσουμε να ρωτήσουμε ίσως το ρόλο. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια απόπειρα, να γράψουν ένα γράμμα οι πρόεδροι και να υποβάλουν οι ομάδες ένα σχέδιο ψηφίσματος, να προσπαθήσουμε να το βάλουμε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την αρχή του ΟΗΕ, σχετικά με την ευθύνη της προστασίας. Η σύσταση είναι της ε, συναδέλφου Μπράτνερ. Ε, συναρμόδια Επιτροπή, η Επιτροπή Ανάπτυξης. Κύριε Μπρέντνερ, έχετε το λόγο. Διαφωτίστε μας. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ε, να σας πω ότι στην ομάδα μας είχε κάνει συζητήσει για το ποιος θα αναλάβει ε, το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσω και τον ε, Μάικλ Κάσμαν από την Επιτροπή ΔΕΒΕ υιοθέτησε το σχετικό κείμενο την προηγούμενη Τρίτη. Πολλά σημαντικά στοιχεία συμπεριληφθήσαν και θα μας ε, φανούν και εμάς ε, χρήσιμα τώρα επί του περιεχομένου. Να σας πω το εξή. Υπάρχει ένα διεθνές πλαίσιο και γίνεται μια συζήτηση ακόμα για την αρχή της ε, ευθύνη της προστασίας. Όπως ξέρετε, υιοθετήθηκε μετά την Γενική Συνέλευση του 2005 η αρχή αυτή και συζητιέται έκτοτε και περνάει από διάφορες ε, φάσεις ανάπτυξης. Ε, καταρχάς, ε, εφαρμόστηκε το 1973 σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Ασφαλείας και την απόφαση του να εφαρμοστεί στη Λιβύη. Αυτή η σύσταση έχει ως στόχο να υπάρξει μια διευκρίνηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι σημαίνει η ευθύνη για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ε, ποιος είναι ο ρόλος μας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της αρχής αυτής. Θα θέλαμε λοιπόν να οριστεί μια διαδικασία να ξεκινήσει μια διαδικασία διαχασμικής συζήτησης προκειμένου να καταλήξουμε σε διευκρινήσεις, σαφήνεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της αρχής αυτής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι καλό θα είναι να υπάρχει μια κοινή, ένας κοινός ορισμός της αρχής αυτής γιατί ως τώρα είναι πολύ αμφιλεγόμενες οι σχετικές συζητήσεις και καθόδεις σε πολλές περιπτώσεις, δεν συμφωνούμε. Νομίζω ότι θα ήθελα η σύσταση να παραμείνει σύντομη, γιατί δεν θέλω να προκαταλάβω τα αποτελέσματα μιας τέτοια διαδικασίας. Θέλω απλά να ξεκινήσει μια διαδικασία και όχι να α, πω εκ των προτέρων ποια θα πρέπει να είναι τα αποτελέσματα της συζήτησης αυτής και θέλω να συνδράμουμε και στην διεθνή συζήτηση. Θα ήταν νομίζω χρήσιμο να υπάρχει μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου επικοδομητικά να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και στην διεθνή συζήτηση και στις διεθνείς εξελίξεις. Άρα, του, του λεχθέντος, η σύσταση αυτή είναι συνοπτική και σύντομη και αναφέρεται στο τι σημαίνει αυτή η ευθύνη, αναφέρεται στους ε, τρεις πυλώνες, σε ό,τι αφορά τη διεθνή αρρωγή της ευθύνης του κράτους και αν αποτύχουν όλα τα υπόλοιπα στην έγκαιρη αποφασιστική αντίδραση καθώς και το ότι περιλαμβάνει τις, ευθύνες, ε, τις πτυχές της ευθύνης πρόληψης, της ευθύνης αντίδρασης και της ευθύνης αναδόμησης. Επίσης, ότι περιλαμβάνει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ότι ασφαλώς η όλη διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τους ε, παράγοντες της ε, κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, ζητούμε από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να συνεχίσει να προασπίζει την αρχή της ευθύνης προστασίας. Αυτά λοιπόν λίγο πολύ περιλαμβάνει η σύσταση και ασφαλώς όλοι έχουμε μία άποψη για το τι θα πρέπει να σημαίνει αυτή η αρχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην παρούσα φάση θέλω απλά να ξεκινήσω μια διαδικασία παρά να δώσω απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ και ανυπομονώ να ακούσω και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατανοώ πλήρως την προσπάθεια την οποία έκανε η κυρία Μπράντερ και θα ήθελα να κάνω κάποια μικρά σχόλια ως εξή. Υπάρχουν τρεις τομείς θα έλεγα που μας ενδιαφέρουν σε σχέση με το θέμα αυτό της σύνδρομης. Θα προσπαθήσω να τα παρουσιάσω κάπως συνοπτικά. Πρώτον, αυτό που έχει σημασία είναι να υπενθυμίσουμε ότι βασικός και μοναδικός στόχος της στρατιωτικής παρέμβασης σύμφωνα με τον τρίτο πυλώνα είναι να αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί πληθυσμοί. Καμία άλλη πρόταση όπως ε, διάφορες αξίες ή κάποιο πολιτικό σύστημα η υποστήριξη της εδαφικής ακαιρεότητας ε, θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν νόμιμα θα έλεγα κίνητρα και αιτιολογήσεις παρέμβασης στρατιωτικής. Με άλλους τρόπους ίσως, αλλά όχι μέσω αυτού που μας ενδιαφέρει. Τώρα δεύτερον, το θέμα είναι η ευθύνη προστασίας, έτσι ονοματίζεται αν θέλετε. Αυτό το έχει λάβει υπόψη της η κυρία Μπραντνερ ε, θυμίζω ότι θα πρέπει σε αυτή την πρωτοβουλία να στρέψουμε την προσοχή μας με πάρα πολύ ε, επιφυλακτικότητα. Ε, στόχος μας είναι να πείσουμε ορισμένες χώρες, όπως η BRICS σαν παράδειγμα, να αναλάβουν την δική τους ευθύνη για προστασία. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, να δοθεί νομική ευθύνη και υπόσταση σε διεθνές επίπεδο, σε αυτή την ευθύνη προστασίας για να υπάρξουν σωστές διεθνείς σχέσεις. Και το τρίτο θέμα είναι το συγκεκριμένο εμπόδιο το οποίο τίθεται σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος αρνησικερίας από πλευράς των μονίμων μελών των, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εγώ θα ήθελα να καταθέσω μια τροπολογία μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να υιοθετήσουν έναν κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος σε εθαλοντικό επίπεδο, μιας και πρόκειται για μόνιμα μέλη, ε, εθελοντικά περιορίζουν το δικαίωμα της χρήσης της αρνησικυρίας στις περιπτώσεις όπου δεν διακινδυνεύεται μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Ευχαριστώ Πρόεδρε εξ ονόματος της κυρίας Νίνσκι, η οποία είναι σκιώδης εισηγήτρια από πλευράς της πολιτικής μας ομάδας, θα ήθελα να μοιραστούμε ορισμένες σκέψεις γύρω από την πρόταση την οποία κάνει η κυρία Μπραντνερ προς την οποία θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης για την ευθύνη προστασίας. Πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια η οποία υποστηρίχθηκε από το διαβημένο Προεδρείο της Επιτροπής μας ομόφωνα. Βασικός στόχος της κυρίας ε, Μπραντνερ, με τον οποίο συμφωνούμε, δεν είναι να ξεκινήσουμε μόνο μια ιδεολογική θεωρητική συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή της αρχής της Εθνής προστασίας, αλλά να βρούμε πρακτικούς τρόπους ε, που μπορεί να λάβει πρακτικές μορφές που μπορεί να λάβει η συγκεκριμένη αυτή έννοια ε, μετά από την πρώτη απόφαση γύρω από αυτό που είχε ληφθεί ήδη το 2005. Πιστεύουμε ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής γύρω από την ευθύνη προστασίας θα πρέπει να στραφεί σε μια δημιουργία μέτρων που θα ονόμαζα προληπτικά. Ε, γνωρίζουμε απαράδεκτες καταστάσεις γενοκτονίας, εθνοκάθαρσης, εγκλημάτων εις βάρος της ανθρωπότητας, γενικά μια σειρά ε, καταστάσεων που μας πείθουν ότι υπάρχει ανάγκη ε, να τεθεί σε εφαρμογή η βασική αυτή αρχή της ευθύνης προστασίας μέσω συγκεκριμένων μέτρων. Όπως είπε άλλωστε και ο κύριος Μενέντες Δεβάγια και θα συμφωνήσω, θα υπογραμμίσω κι εγώ, ότι η αρχή αυτή της ευθύνη προστασίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ε, με, ε, κάποια πρόφαση, υπό τη μορφή πρόφασης έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται στρατιωτικά μέσα και να υπάρχουν στρατιωτικές παρεμβάσεις. Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να θέσει σε λειτουργία μια, μια ενδιαφέρουσα σειρά πρωτοβουλειών προληπτικής φύσεως. Μια άλλη πλευρά την οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω σε σχέση με αυτήν την σύσταση προς το Συμβούλιο είναι να μην να μείνουμε ε, θα έλεγα εσωστρεφείς. Προφανώς θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να προκαλέσουμε την έκφραση αλληλεγγύης των κρατών μελών, αλλά και των υπολείπων περιφερειακών οργανώσεων. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια δράση προς την ακινητοποίηση αυτή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τελειώσω ευχαριστώντας για μια ακόμη φορά για την κυρία Μπραντνερ για την έκθεσή της και να επιμείνω όπως είπε και η κυρία Νίνσκι εξ ονόμαστος της οποίας ε, ομιλώ να μην ε, παραποιηθεί η αρχή και η μορφή της συγκεκριμένης αυτής ιδέας από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό τρόπο να μπορέσει να καταλήξει σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα θέσουν σε εφαρμογή την ίδια αυτή αρχή. Πρόεδρε. Χαίρομαι για την έκθεση της κυρίας Μπράτνερ, η οποία αναφέρεται σε ένα πρόβλημα που μας απασχολεί διαρκώς και στο οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση τώρα η διεθνής κοινότητα. Θα υποστήριξω τα όσα μας πρότεινε ήδη ο κύριος Μέντες Δεβάγε, τις τροπολογίες, διότι στην πρώτη ανάγνωση της εκθέσεως αυτής, εγώ διαγνώσκω μια απουσία ισορροπίας μεταξύ του πρώτου τμήματος της αιτιολογικής σκέψης που είναι πολύ αναλυτική και αναφέρεται σε πραγματικά προβλήματα. Στο σημείο Z, παραδείγματι, G σε σχέση με τις εντάσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και άλλων μορφών διαμεσολάβησης, θέματα που είναι πολύ πολιτικά δηλαδή, αφενός αφετέρου δε τις στάσεις στα σημεία 1, 2, 3, 4 και 5, όπου γίνεται λόγος για ομάδες, συναντήσεις, εκθέσεις και το καθεξής. Άρα, δεν βλέπω πώς αυτή τη στιγμή αλλά θα το δούμε πιστεύω στην πορεία με τις τροπολογίες πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις με τις σε αυτές τα προβλήματα που έχουμε. Ναι, πρέπει να διευκρινίσουμε τις έννοιες, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα στην υλοποίηση, όπως λέει και ο κύριος Ολαφράγκα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής αλλά πρέπει νομίζω να ε, διατυπώσουμε συστάσεις με πολύ πιο σαφές μήνυμα. Γι' αυτό και υποστηρίζω τις συστάσεις πολύ έντονα πολιτικού χαρακτήρα του κύριου Δευναία. Χρειάζεται λοιπόν επαναδιατύπωση το έγγραφο αυτό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπράντερ που ανέλαβε να το, κάνουμε, να το συνεχίσουμε την κυρία Μπρέτπουλς. Αλλά θέλει ακόμα πολύ δουλειά. Ευχαριστώ κυρία Νέιτς. Ε, Πρόεδρε, συνάδελφοι, επειδή δεν είναι εδώ η τη συζήτρια κυρία ΠΕΚΑ, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης που μας ε, υπέβαλε η Φραντσέσκα. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία σε πρώτη φάση να εμβαθύνουμε πραγματικά την αρχή της ευθύνης προστασίας και να διευκρινίσουμε τι εννοούμε για μια σύντομη χρονική περίοδο φαινόταν ότι η ευθύνη προστασίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει επεμβάσεις, παρεμβάσεις σε ξένες χώρες. Οι αντιδράσεις στην παρέμβαση στη Λιβύη και κυρίως μετά την παρέμβαση αυτά που έγιναν κατέδειξαν ότι τα πράγματα ήταν πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι εκ πρώτη όψεω φαινόταν. Δεν ξέρω τι είδου τροπολογίε θα καταθέσουμε. Κατά πάσα πιθανότητα όμω έχω την αίσθηση ότι θα είναι απαραίτητο να επιμείνουμε στη σημασία των δύο πρώτων σταδίων της ευθύνης ε, της ε, προστασίας και να μην περάσουμε κατευθείαν στο τρίτο στάδιο. Ακόμα και αν η διεθνής κοινότητα ήθελε και μπορούσε σε κάθε περίπτωση να αντιδρά συλλογικά και να παρεμβαίνει οποτεδήποτε υπήρξε, υπάρχει τέτοια μεταχείριση των πολιτών από, τους, από τις κυβερνήσεις και επίσης να έχουμε υπόψη ότι η ευθύνη της προστασίας περιλαμβάνει και την ευθύνη αναδόμησης ενός κράτους, το οποίο κατεστράφτη σε πρώτη φάση και αυτό που μάθαμε, ή εν πάση αυτό που θα έπρεπε να έχουμε μάθει τα τελευταία 20 χρόνια, είναι ότι η αναδόμηση, η δόμηση ενός κράτους μετά την ε, κατάρρευσή του, μετά την καταστροφή του, καταναλώνει πολύ πιο πολύ χρήματα, πολύ πιο πολύ χρόνο και πολύ πιο πολύ κόπο από ό,τι πίστευα. Και ας δούμε τι γίνεται στη δικιά μας τη γειτονιά, στη Βοσνία Ζεγοβίνη, στο Κόσοβο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι δύο χώρες αυτές σήμερα βρίσκονται στην άριστη κατάσταση, γιατί δεν βρίσκονται. και απέχουν μόνο 500 έως 1000 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα όταν η κατάσταση είναι και ακόμα χειρότερη από αυτή που γνωρίσαμε εκεί, στη Βοσνία Ζερβοβίνη, στο Κωσυφοπαίδιο. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει αυτό το σχέδιο σύστασης γιατί μας ε, καλεί να εξετάσουμε τις ενδεχόμενες συνέπειες της αρχής αυτή. Ασφαλώς δεν πρόκειται να περιλάβει όλα τα θέματα που αφορούν την ε, διεθνή αντίδραση. Εγώ σε ό,τι αφορά την δυνατότητα να παρέμβουμε σε οποιαδήποτε φάση που υποφέρουν πολίτες, ορίζω τη σύσταση αυτή, όπως σας είπα και θα δούμε κατά πόσο θα καταθέσουμε τροπολογίες, αλλά θεωρώ ότι θέτει τη βάση για το μελλοντικό μας έργο και για ένα καλό έργο μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκόμες, ευχαριστώ πρόεδρα και εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Φραντσέσκα Μπράβνερ για την πολύ χρήσιμη αυτή έκθεση. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε να ξεκινήσει η συζήτηση στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα, είναι το διακύβευμα στην παρούσα φάση, δεν είναι το να κάνουμε κάποιες μεγάλες δηλώσεις, ούτε να νομιμοποιήσουμε την παρέμβαση σε διάφορες περιοχές στον κόσμο. Το θέμα είναι να νομιμοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε το νομικό πλαίσιο εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων, έτσι ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε όπου αυτό είναι απαραίτητο και όπου χρειάζεται. Υπάρχουν περιοχές που χρειάζεται για να σταματήσουν γενοκτονίες, για να σταματήσουν μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και εγκλήματα πολέμου. Παράδειγμα η Ρουάντα η Σρεμπρένιτσα. Λοιπόν, έστω και τώρα, εάν δεν υπάρχει νομική δυνατότητα για να σταματήσουμε τις παραβιάσεις, είναι σαφές ότι θα συνεχίσουν οι παράνομες αυτές ενέργειες, όπως άλλωστε το βλέπουμε στη Συρία γιατί στη Συρία υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παρεμβαίνουν και προς την κατεύθυνση αυτή και που προκαλούν περαιτέρω παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκαλούν περισσότερα εγκλήματα πολέμου κτλ. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με την ανάγνωση που κάνετε για την βραζιλιάνικη πρόταση. Προφανώς έχει σημασία να ορίσουμε τα όρια αυτής της νομικής ευθύνης κατά τη διάρκεια της προστασίας, της άσκησης της προστασίας. Το θέμα είναι όμως να δούμε πού βρίσκεται το επίπεδο προστασίας το οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Πρώτον, θα πρέπει να έχουμε κάποιον, και αυτός ο κάποιος θα πρέπει να είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο θα λέγει ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η στρατιωτική παρέμβαση πρέπει να υπάρξει, είναι θεμητή και απαραίτητη για να σταματήσουν οι σκοτομοί. Πριν λοιπόν ορίσουμε το συγκεκριμένο θέμα της ευθύνης κατά τη διάρκεια της προστασίας, Γνωρίζω πολύ καλά ε, το τι υποστηρίζει η Βραζιλία. Ξέρω ότι η Βραζιλία ε, δεν ε, συμφώνησε με αυτό που έγινε στη Λιβύη. Εγώ διαφωνώ με τη Βραζιλία. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν λάθος το ότι σταματήσαμε τη σφαγή στη Βεγγάζη. Εγώ πήγα εκεί και είδα. Εγώ δεν υπερασπίζουμε την πολιτική μου οικογένεια. Ήταν σωστό να προχωρήσουμε στο να σταματήσει αυτή η σφαγή γιατί 20 λεπτά αργότερα να είχαμε παρέμβει θα είχαμε ξανά τη Ρουάντα και τη Σβεμπρένιτσα στην Πεγκάζη. Συνεπώς λοιπόν θέλω η παρέμβαση αυτή να γίνεται με τρόπο ο οποίος να είναι διακανονισμένος και δεν μπορεί να γίνει αυτό στην παρούσα φάση. Πρέπει λοιπόν εδώ να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εγώ δεν θέλω να γίνονται παράνομες ε, ενέργειες. Το σωστό όργανο, το κατάλληλο όργανο είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν εκεί αφού προχωρήσουμε σε μια τέτοια ρύθμιση να περάσουμε στις ανησυχίες της Βραζιλίας. Πολλοί πιστεύουν στον κόσμο σήμερα ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν είναι νόμιμο σε εισαγωγικά, δεν νομιμοποιείται να λαμβάνει αποφάσεις. Και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς συνεχίζουμε το ερώτημα αυτό να το αποκρύβουμε. Δεν θέλουμε να συζητάμε, ε, θα πρέπει εμείς να ζητήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε μία μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας παράλληλα να ακολουθήσουμε μία στάση επιρροής όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξει περιορισμός της άσκησης του δικαιώματος αρνησικυρίας από πλευρά των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό είναι απαραίτητο. Νομίζω λοιπόν ότι οι προτάσεις της κυρίας Μπραντνερ της Φραντσίσκα Μπράτνερ θα οδηγήσουν σε μια συνενετική λύση, μια λύση η οποία θα περιλαμβάνει το ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν θα χρησιμοποιούν απεριόριστα το δικαίωμα βέτο εφόσον τίθενται θέματα ασφάλειας πληθυσμών κτλ. Ε, Mr. Tannock. Κύριε πρόεδρε, Είναι πολύ θαραλέα η κυρία Γκόμες όταν ε, αντιτίθεται στις θέσεις της κυβέρνησης της Βραζιλίας και της αντιπολίτευσης. Εγώ θα πω ότι θα υποστηρίξω την πρόταση ώστε και η Γαλλία και η Γερμανία και η Βραζιλία να είναι χώρες ε, χωρίς δικαίωμα του ΝΑΤΟ, μόνιμα μέλη όμως στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και υπάρχει, όπως είπαμε, ήδη η έννοια του δικαιώματος στην προστασία, right to protect, αντί για την ευθύνη. Έχει ξεκινήσει από την περίοδο του πολέμου στο Ιράκ. Είναι πολύ πιο εύστοχος όρος δικαίωμα για προστασία. Και όταν χώρες όπως η Κίνα αντικείται σε κάθε έννοια επέμβαση στο εσωτερικό άλλης χώρας, ε, έχουμε αποτελέσματα όπω αυτά που βλέπουμε τώρα στη Συρία. Η ευθύνη όμως, η υπευθυνότητα, η υποχρέωση ακόμη που σηματοδοτεί η δεύτερη έκφραση responsibility to protect δεν δίνουν την ευρύτερη ε, εικόνα δεν εκφράζουν την ευρύτερη υποχρέωση και για την ανοικοδόμηση μιας χώρας μετά την καταστροφή. Γιατί μην ξεχνάμε σε σχέση με τη Βόρεια ε, Κορέα που τους μολι μόλις τώρα. Ύστερα από 30-40 χρόνια όλα τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί ε, και ακόμα και στην Ερυθρέα ή τη Συρία μέχρι τώρα κανείς δεν φανταζόταν θα μπορούσε να υπάρξει επέμβαση από το εξωτερικό γιατί ε, κάποιες ε, περιπτώσεις, κάποιες καταστάσεις μπορεί να θεωρηθούν πολύ ε, επικίνδυνες και να μην αποτολμήσει κανείς να ε, επέμβει. Εγώ προσωπικώς για το Ιράκ είχα υποστηρίξει την επέμβαση, αλλά τώρα με δεδομένα τα όσα ήδη γνωρίζουμε δεν είμαι σίγουρος ότι θα το έπρατα. Πρέπει όμως με όσες καλές προθέσεις ε, σε μια αρχική ε, παρέμβαση να αποτρέπονται πάντα οι θάνατοι αθώων. Ίσως λοιπόν κάποιοι συνάδελφοι να θέλουν να περιοριστούν τα δικαιώματα της αρνησικηρίας για χώρες όπως η δική μου, ακόμα και σε θέματα ιερά όπως είναι αυτό της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε πόσο περίπλοκες είναι οι στην ε, εξωτερική πολιτική και πόσο λεπτές ισορροπίες και στάθμιση εθνικού, ευρωπαϊκού, συμφέροντος ανθρωπινών δικαιωμάτων, εμπορικών οικονομικών σχέσεων. Ας δούμε τι κάνουμε σε σχέση με την Κίνα, παράδειγμα τη δηλαδή, λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, που έχει επέμβει στο Θιβέτ με πολύ δυσάρεστες εξελίξεις, αλλά κανείς δεν τολμάει να αντιταχθεί σε αυτήν. Ευχαριστώ κυρία Μπράτνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας προσφέρετε να σχολιάσουμε την πρόταση αυτή. Βεβαίως ε, εμείς θέλουμε να επιμείνει στο θέμα της ευθύνης για προστασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο μια συγκεκριμένη έκθεση, αλλά και με τις τακτικές αιτήσει ε, συστάσεις του προς το Συμβούλιο, εν ώψη και της ε, ε, γενική συνέλευση. Πάντοτε υπογραμμίστε την ανάγκη, την ευθύνη για προστασία, αλλά έχετε και πολύ σημαντικέ εκδηλώσεις διοργανώσει. Πρέπει να συζητείτε το θέμα αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από την η διαδικασία έγκριση αυτής της έννοια που είναι πολιτική και όχι νομική, έχει εξακολουθήσει να υπερασπίζεται την διατύπωση του 2005, επιδιώκοντας μια καλύτερη συνεννόηση για το τι σημαίνει αυτή, ιδιαίτερα με τις συζητήσεις που έχουν γίνει στα Ηνωμένα Έθνη, το ρόλο των διεθνών οργανισμών, στους οποίους περιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μία συζήτηση που, έγινε, που ξεκίνησε από πέρσι για τον τρίτο πυλώνα που έχει και το στρατιωτικό σκέλος και μπορεί να οδηγήσει σε δύσκολε αποφάσεις. Εκεί πέρα εντάσσεται και η ε, επίλυση των διαφορών και η διπλωματία. Έχει πάει καλά αυτή η συζήτηση μέχρι τώρα, αλλά ε, ενδεχομένω να δούμε εξελίξει σχέση με τι χώρε του Νότου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ζητεί να εστιαστούμε περισσότερο στην πρόληψη ή την αποτροπή και γι' αυτό στην επόμενη έκθεση του Γενικού Γραμματέου περιμένουμε ε, να εκδοθεί και εν ώψη ελληνική συνελεύσεω. Πιστεύω ότι θα αποτελέσει μια ευκαιρία να εστιαστούμε στην ε, ιδέα αυτή και να σταθμίσουμε πολύ πιο ισότιμα τις ε, προσεγγίσεις και το τελικό κομμάτι του τρίτου πυλώνα ως προς την παρέμβαση. Ασφαλώς. Και θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στη διατύπωση της εκθέσεως ε, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις υπόλοιπες χώρες, ιδιαίτερα με τον Νότο. Θεωρούμε ευπρόσδεκτη τη συμβολή της Βραζιλίας στον δημόσιο διάλογο και ίσως κάποια κράτη-μέλη διαφοροποιούνται σε σχέση με τις συστάσεις. Ένα κρίσιμο σημείο είναι ότι χρειάζεται διεξοδική συζήτηση και προαγωγή της ιδέας αυτής της ευθύνης για προστασία, χωρίς όμως να χαρακτηρίζεται αποκλειστικά ως μια πρόταση ή ιδέα ή έννοια που εκφράζει μόνο τα δυτικά κράτη. Πρέπει και οι εταίροι από τον Νότο και δεδομένων των ε, ιδιαιτεροτήτων και της επέμβασης στη Λιβύη να ε, εμπλακούν σε αυτήν την ιστορία. Υποχρέωση λοιπόν για ανάληψη και συνεργασίε σε τη σχέση με τρίτες χώρες για να μπορέσουμε να συστήσουμε πιο αναλυτικά την αρχή τη ευθύνη για ε, προστασία. Και εδώ δεν μπορούμε να λησμονούμε φυσικά και όλε τι έννοιες του ανθρωπιστικού δικαίου. Οι συνθήκε τη Γενέβης ε, φυσικά ε, ισχύουν εφόσον έχουν κυρωθεί όμως οι δικασίες καμιά φορά είναι περίπλοκες και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση όταν συζητούμε νέες έννοιες όπως την ευθύνη για προστασία γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με επιλογές νομικού τύπου, ένομου τύπου δηλαδή από πλευράς των κρατών με συνέπειες. Κυρία Μπράτντερ. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλιά σας. Συνάδελφοι, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση και νομίζω ότι αυτό που βασικά αποκομίζω από τη συζήτηση αυτή είναι ότι εσείς ως συνάδελφοι και ως πολιτικές ομάδες θέλετε να, να διατυπωθούν συστάσεις για το πώς θα θέλαμε εμείς να εφαρμοστεί η αρχή αυτή και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Ως τώρα, εγώ η ίδια δεν ε, διατύπωσα συστάση, αλλά και από την κυρία Νένσκι ε, μας μίλησε για τις πρακτικές εφαρμογές ε, της, εφαρμογής της αρχής ε, και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και η κυρία Νέιτς και η κυρία Γκόμες και οι υπόλοιποι συνάδελφοι κάναν κάποιες προτάσεις σχετικέ. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθώ λοιπόν και θα είναι πολύ πιο δύσκολες οι συζητήσεις στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται. Συμφωνώ ιδιαίτερος με την κυρία Νένσκι και τον κύριο Σολανφράγκα ότι το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί η αρχή αυτή και τι σημαίνει για την καθημερινή μας πολιτική, για τις καθημερινές πολιτικές μας. Ποια είναι η ευθύνη μας για να αποτρέψουμε γενοκτονίες. Έχουμε τα εργαλεία που χρειάζεται. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που είναι σημαντικά και πρέπει να τα απαντήσουμε. Όπως μιλήσατε επίσης για προληπτικά εργαλεία, προληπτικά μέσα. Βασικό και αυτό. Αν θέλουμε να είναι αξιόπιστη η διαδικασία αυτή και όχι να αποτελεί μια δικαιολογία για στρατιωτική επέμβαση. Και ύστερα ο κύριος Μενεζεβάια είπε ότι πρόκειται για πρόληψη γενοκτονιών και πολύ συγκεκριμένες ε, ανθρωπιστικές ε, καταστροφές. Συμφωνώ. Και σε ό,τι αφορά το Μάλι, για παράδειγμα, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαρη, να μην μπλέκουμε δύο ειδών καταστάσεις. Χάρηκα λοιπόν για το σχόλιο αυτό που κάνατε και σε περίπτωση που καταθέσατε σχετικέ σχετικές για να το διευκρινίσετε περαιτέρω το θέμα αυτό, θα χαρώ να τη συμπεριλάβω. Αυτό που είπε ο κύριο Σαλαφράγκα για το ότι θα πρέπει να, δράμε, να δρούμε από κοινό με τις, άλλες, ε, φορεί και όχι από μόνοι μας. Ναι, φυσικά, σε συνεργασία και με του άλλου περιφερειακού φορεί με την, ε, τον Αραβικό Σύνδεσμο, με την Αφρικανική Ένωση. Βεβαίως και η κυρία Ντεκάιζερ και η κυρία Γκόμες, είπατε ότι οι απαντήσεις δεν είναι οι σωστές απαντήσεις για το ύψος και το μέγεθος του προβλήματος. Κοιτάξτε, ε, αν θέλετε, εμείς ως Κοινοβούλιο να δώσουμε ήδη τις δικές μας απαντήσεις στα πλαίσια του διαθεσμικού διαλόγου, θα χαρώ να τις υποβάλω, να κάνω και εγώ κάποιες προτάσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συζήτηση και προσβλέπω στις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εκτός μικροφώνου, μάλιστα, την, την 5η 12 η ώρα η προθεσμία για την καταθέση τροπολογιών. Μάλιστα, και τώρα περνάμε το 6 της ε, ημερήσιας διάταξη. πρόταση ψηφίσματο σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο συνάδελφος Χάουιτ είναι ο εισηγητή. Έχετε το λόγο, τροπολογίε μέχρι τις 28 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα. Αυτή ήταν η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω αναφερόμενο στην πρόσφατη επίσκεψή μου στη συγκεκριμένη χώρα πριν μια εβδομάδα. Λόγω και της πολιτικής κρίσης η οποία σοβεί στη χώρα, με συγκεκριμένα βία γεγονότα στις 24 Δεκεμβρίου οδήγησε στην έξοδο ορισμένων κοινοβουλευτικών από την συνέλευση, την εθνοσυνέλευση στα Σκόπια. Υπήρξαν γενικά βίες αντιπαραθέσεις. Το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης εγκατέλειψε την Εθνοσυνέλευση και απειλεί να σαμποτάρει τις δημοτικές εκλογές που προβλέπονται για τον μήνα Μάρτιο. Αυτά είναι συμβάντα καθόλου επιθυμητά. Το είπαμε αυτό και εμείς και ο Επίτροπος και τα κράτη-μέλη προσπαθήσαμε να επηρεάσουμε τα πράγματα, να κάνουμε δηλώσεις έτσι ώστε να λύσουμε τα αντιπαρατηθέμενα μέρη, να ξεπεράσουν τις διαφορές τους Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος. Εγώ συναντήθηκα με όλα τα πολιτικά κόμματα και ιδιωτικά και δημόσια. Οι συναντήσεις ήταν επικοδομητικές. Αποφάσισα να δημοποιήσω αρκετές από τις πληροφορίες που συνέλεξα, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Και θα ήθελα να μεταφέρω αυτές τις πληροφορίες να πω ότι λυπάμαι για την σημερινή πολιτική κατάσταση η οποία θέτει σε αμφισβήτηση τη μελλοντική πρόοδο της χώρας. Ζήτησα από τα κόμματα με τα οποία συναντήθηκα να κάνουν βήματα προόδου. να σεβαστούν τις αποφάσεις που είχαν λάβει στο παρελθόν. Πράγματι η πολιτική της χώρας μου είχαν πει ότι είχε υπάρξει και μια κάποια θετική όθηση και σε σχέση με το θέμα του ονόματος. Και δεν θα πρέπει λόγω της κρίσεως να σταματήσει η όθηση αυτή. Νομίζω ότι τον Ιούνιο υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία για να υπάρξει μια θετική απόφαση αλλά αν οι εξελίξεις στη συγκεκριμένη χώρα τις επόμενες ημέρες αποτρέψουν να σημειωθεί κάποια πρόοδος, αυτό δυστυχώς μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις ε, ε, για την επίλυση των προβλημάτων, ε, δυστυχώς. Είπα ήδη ότι σε σχέση με αυτά τα οποία συνέβησαν την 24η Δεκεμβρίου είναι θέματα που δημιουργούν ερωτήσεις, ερωτηματικά σε σχέση με τις δημοκρατικές δομές της χώρας και τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει σε αμφισβήτηση την στήριξη προς την χώρα αυτή και στον τομέα των πολιτικών θεσμών και δημοκρατικών δομών και νομίζω ότι οι διαφορές μπορεί να επιληθούν. Είπα επίσης, και αυτό χωρίς καμία ευχαρίστηση, ότι αν δεν επιληθεί η παρούσα κρίση, και εγώ μάλιστα έκανα την πρότασή μου και επίσημα, ο κύριε Μπροκ, το Κοινοβούλιο να αναβάλει την ψηφοφορία της στην Επιτροπή μας, η οποία θα πρέπει να γίνει σε λίγες εβδομάδες για την έκθεσή μου. Το λέγω αυτό γιατί νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει μια έκθεση η οποία να περιλαμβάνει θετική σύσταση για την ένταξη της χώρας και πιστεύω ότι όμως λόγω της σημερινής κατάστασης στη συγκεκριμένη χώρα είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε μια αρνητική έκθεση και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να δω. Ελπίζω λοιπόν ότι μια αναβολή της ε, έκθεσής μας ε, θα είναι μια προειδοποίηση προς τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Εμείς θέλουμε να ξεπεράσει η χώρα τα πολιτικά της προβλήματα, την πολιτική κρίση. Εδώ να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές με τους οποίους διαβουλεύτηκα. Ε, συναντήθηκα μαζί τους και πριν πάω στα Σκόπια και τους εκπροσώπους των Πρασίνων της Γκουε, ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και όλοι υποστηρίζουν την πρόταση αναβολή την οποία σας κατέθεσα επίσημα σήμερα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό και νομίζω ότι η ενότητα των θέσεών μας απέναντι στα συγκεκριμένα προβλήματα θα βοηθήσει να ξεπεραστούν τα προβλήματα στα Σκόπια. Πρόεδρε, θα ήθελα εγώ να σχολιάσω κάποιες από τις τροπολογίες και να ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων. Εγώ με την στήριξη της γραμματείας θέλω να συνεχίσω τις διαπραγματεύσεις αύριο για συμβιβαστικές προτάσεις έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι, έτσι ώστε αν υπάρξουν κάποια βήματα προόδου στη χώρα αυτή να προχωρήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες, δεν μπορώ να τα σχολιάσω, να αντισχολιάσω κάθε μία ξεχωριστά. Προσπάθησα να τις ομαδοποιήσω όσο καλύτερα μπορούσα, να πω ότι για την 7 των Πασίνων σχετικά με το θέμα του ονόματος ε, ζητά να επιληθεί πριν το τέλος των διαπραγματεύσεων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, μία πρόταση λίγο διαφορετική. Θα ήθελα να εμείνουμε πιο κοντά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τις εννέα ε, τροπολογίες στο Γιανόφ σχετικά με τις βουλγαρικές θέσεις. Κοιτάξτε, ε, εννέα αιτιολογικές σκέψεις από τις 16 να αναφέρονται στη Βουλγαρία είναι κάτι το υπερβολικό. Το θέμα της, το γλωσσικό είναι κάτι θα έλεγα σημαντικό, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο επικοδομητικοί στις προτάσεις τροπολόγησης. Γι' αυτό να πω σε πολλά άλλα μέλη από τη Βουλγαρία τα, με τα οποία συναντήθηκα. Θα ήθελα να πω ότι ε, θα συμφωνήσω μαζί τους με επικοδομητικό τρόπο να βρούμε κάποιες συμβιβαστικές λύσεις με τις οποίες θα ικανοποιούνται κάποιες από τις ε, θεμητές ανησυχίες τους και δεν θα θέσουμε σε αμφισβήτηση την σύνολη ισορροπία της έκθεσης. Για την παράγραφο 1, ενθυμίστε πέρυσι, είχα συστήσει να υπάρξει μια σαφής δήλωση του Κοινοβουλίου για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και αυτή παραμένει πάντα η ελπίδα μου. Πάρα πολλά μέλη λόγω της σημερινής κατάστασης θέλησαν να τροπολογηθεί το πρώτο άρθρο. Και αυτό ακριβώς δείχνει την ανάγκη που υπάρχει να υπάρξει μια αναβολή. Θα ήθελα εδώ λοιπόν να πω ότι κατανοώ τα μέλη, 26 θα έλεγα, η τροπολογία 26 μπορεί να συνδυαστεί με την δική μου 36 και μπορεί να υποστηριχθεί σχετικά με το θέμα των σχέσεων καλής γειτονίας έχουν κατατεθεί πάρα πολλές τροπολογίες 29, 32, 34, 35, 38 της κυρίας Κοπάν ακούσαμε καλά. Ε, νομίζω ότι υπάρχει διαφορετική διατύπωση με την 41 αλλά νομίζω ότι λέμε τα ίδια πράγματα και θα μπορέσουμε ε, σε δύο παραγράφους να συνδυάσουμε με μια συμβιβαστική πρόταση τα προβλήματα. Για την παράγραφο 3 οι λέξεις game changer ε, δεν την προτιμούν κάποια μέλη. Θα δω ακριβώς τι μπορώ να κάνω για να αλλάξω τη διατύπωση σχετικά με τον διάλογο τον ενταξιακό υψηλού επίπεδου και την τροπολογία 50 είναι σαφές ότι μέχρι τώρα έχουν υπάρξει κάποιοι στόχοι οι οποίοι έχουν επιτευχθεί. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, να δείξουμε την προσπάθεια που έκανε η συγκεκριμένη χώρα. Τώρα, για την τροπολογία των πρασίνων της κυρίας Κορνέλησεν, κατανοώ με την διαδικασία αυτή, αλλά δεν ξέρω νομικά τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με το greening αν ακούσαμε. Τώρα, έχουν κατατεθεί πάρα πολλές τροπολογίες από όλες τις μεγάλες πολιτικές ομάδες. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Ελπίζουμε η κατάσταση στη χώρα να μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε μια διαφορετικό ε, ε, αποτέλεσμα. Τώρα για το θέμα της κατάργησης των θεωρήσεων, 69 τροπολογία κτλ. Θα συμφωνήσουμε για να διατηρηθεί το καθεστώς αυτό, ήταν κάτι το πάρα πολύ θετικό για τη χώρα. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες τις οποίες θα μπορούσα να δεχτώ. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο όμως είναι να υπάρξει πολιτική ουδετερότητα On multi-ethnic education, Νομίζω ότι στην κριτική την οποία κάνω και στην δική μου έκθεση σε διάφορους τομείς της εσωτερικής πολιτικής θα υπάρξει συμφωνία για, το διεθνές, για την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που ίσχυε πέρυσι. Δεν ξέρω αν η διατύπωση η οποία προτείνεται στην παρούσα φάση είναι πράγματι επικοδομητική αλλά νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές τροπολογίες για τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα που θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά. Θα οδηγηθούμε νομίζω σε μια συνενετική διατύπωση. Υπόσχομαι στους Έλληνες συναδέλφους αυτό που υποσχέθηκα και στους Βούλγαρους με επικοδομητικό τρόπο θα σταθώ στις προτάσεις τους. Θα μπορούσα να σας κουράσω ακόμα περισσότερο, αλλά προτιμώ ίσως να απαντήσω σε συναδέλφους οι οποίοι μπορεί να θέσουν τα θέματα τους. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις. Το κόμμα της αντιπολίτευσης είχε το συνέδριό του, δεν έχει αλλάξει την θέση του, απειλεί ακόμα και τώρα να καταθέσουν την παρέτησή τους ε, ε, από την ε, Εθνοσυνέλευση της χώρας την ημέρα των εκλογών και από πλευράς του κόμματος του κυβερνητικού εξεδόθη μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η, προσ... η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων των κομμάτων στις τοπικές εκλογές θα παραταθεί μέχρι το επόμενο Σάββατο το κόμμα της αντιπολίτευσης της αξιωματικής είχε πει να υπάρξει μια συμφωνία για το θέμα αυτό, αλλά για τις εθνικές εκλογές, όχι για τις δημοτικές. Οπότε δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής θέσεων μέχρι τώρα στα μεγάλα κόμματα. Και νομίζω ότι παραμένει ο στόχος της ε, προσπάθειας επίτευξης μιας συνενετικής πρότασης σε σχέση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Αρμόδιο Επίτροπο. Έχουν κάνει προσπάθειες, έχει αναβάλει την επίσκεψή του στα Σκόπια που προεβλέπεται στα πλαίσια του επομένου διαλόγου υψηλού επίπεδου ενταξιακού. Ξέρω ότι είναι σε στενή επικοινωνία και ο ίδιος ο Επίτροπος με τους ηγέτες των δύο μεγάλων κομμάτων και ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος στην αντιμετώπιση της πολιτικής κρίσης στην ΦΥΡΟΜ έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα απαιτούμενα βήματα. Είχα την ελπίδα ότι θα σας έλεγα διαφορετικά πράγματα σήμερα, λυπάμαι όμως, αλλά βρισκόμαστε στην σημερινή κατάσταση. Ελπίζω τα πολιτικά κόμματα, ελπίζω οι πολίτες, η κοινωνία, οι οργανώσεις των πολιτών σε αυτή τη χώρα να κατανοήσουν πόσο σοβαρή είναι η κρίση αυτή, όχι μόνο σε επίπεδο εσωτερικών υποθέσεων, αλλά σε επίπεδο ε, ε, της θέσης της χώρας συνολικά σε διεθνές επίπεδο. Έφτασε η ώρα η χώρα να επανέλθει στο σωστό δρόμο, να ξεπεράσουν τα μικροκομματικά προβλήματα και αυτό θα πρέπει να επιδιωθεί από όλους. Ο Επίτροπος Φούλε έχει ε, εκφράσει την υποστήριξή του στις προσπάθειες ξεπεράσματος της κρίσης και ελπίζω ότι και τα πολιτικά ε, κόμματα και στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να πιέσουν ε, τα κόμματα που ανήκουν στις πολιτικές τους οικογένειες για να δείξουμε ότι εμείς εμπιστευόμεθα τη χώρα αυτή για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη χώρα αυτή ενωμένα ε, και να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Ο κύριος Κουκάν, πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ τον κύριο Χάουιτ, τον συγκητή, για την καλή δουλειά του. Τον υποστηρίζουμε, υποστηρίζουμε την παρουσίαση Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίση όλου του αδέλφου που παρακολουθούν την κατάσταση στη Μακεδονία και που συνεισφέρουν με τις τροπολογίες του στη βελτίωση τη εκθέσεω. Όπως παρακολουθήσαμε, όπω συζητήσαμε και σε προηγούμενη ε, συνεδρίαση, είναι ισορροπημένη έκθεση. Πλην όμως, πλην όμως, μεγάλο όμως, η εσωτερική κατάσταση, η πολιτική κατάσταση στη χώρα είναι πολύ ανησυχητική ακόμη, με εξελίξεις που μπορεί να έχουν συνέπεια για την έκθεση. Πολιτικές δηλώσεις οι οποίες ακολουθούν τα γεγονότα της 24 Δεκεμβρίου δεν μας φέρουν πιο κοντά σε λύση και προσωπικώς φοβούμε ότι η πολιτική βούληση για επικοδομητικό διάλογο δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί. Ανησυχώ για τις εξελίξεις και ιδιαίτερα για την αποχή από τις χειρογραφικές εργασίες από πλευράς αντιπολίτευσης και ε, την ανακοίνωση της αποχής από πλευράς τους πάλι στις δημοτικές εκλογές. Σε μια κατάσταση τέτοια, ε, με μια, ε, μια θετική ή μάλλον ουδέτερη αξιολόγηση της ε, κατάστασης ε, μπορεί να αποδειχθεί προβληματική. Γι' αυτό καλώ όλους τους Μακεδονίτες πολιτικούς να εντατικοποιήσουν το έργο τους, τις προσπάθειές τους για να βρουν λύση στην κατάσταση. Η αποχή δεν είναι λύση, καθώς δε μάλλον μπορεί και να παρεμποδίσει την ε, υλοποίηση των επιτευγμάτων της χώρας και στο βαθμό αυτό τίνω να συμφωνήσω με την πρόταση του εισηγητού για αναβολή της ψηφοφορίας για την έκθεση. Βέβαια πρέπει να προχωρήσω και σε διαβουλεύσεις με την πολιτική μου ομάδα. Η συνεδρίαση συγητού και σκιωδών συγητών έχει προγραμματιστεί. Πιστεύω ότι θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για ε, επίτευξη μια καλής λύση συνενετική για το πώ θα διαμορφωθεί περαιτέρω διαδικασία. Είναι προ το συμφέρον μα, πιστεύω να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία διότι πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποτελέσει, να διαδραματίσει το ρόλο ενός παράγοντα θετικού που θα συμβάλλει στη λύση. Δεν πιστεύω ότι τίθεται να αμφιβόλω η ε, πρόοδοι σε αυτή τη διαδικασία της Μακεδονίας, αλλά δέχεται να παρεμποδιστούν οι περαιτέρω πρόοδοι. Είμαι ε, βέβαιος ότι όλοι οι πολιτικοί της ε, Μακεδονίας θα συμπεριφερθούν κατά τρόπο υπεύθυνο και σοβαρό, αν και ομολογώ πως αυτή μου η ελπίδα σιγά σιγά εξασθενεί. Επίσης για τις συμβαστικές προτάσεις δεν τις έχουμε δει ακόμη. Και θα ήθελα να ακολουθήσουμε τη σύσταση του εισηγητού για την χρήση του όρου «μακεδονικός» μαζί με το φύρο μία φορά τουλάχιστον στην έκθεση. Κατά τα άλλα για τις τροπολογίες προτείνω τα εξή. Δεν υποστηρίζω τις τροπολογίες που θα οδηγούσαν το ή άλλως στην επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα. Δεν σκοπεύω να υποστηρίξω μονομερείς τροπολογίες, τροπολογίες οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ένταση στις σχέσεις ε, με τη Βουλγαρία ή με την Ελλάδα και εν τέλει φρονώ ότι παρά το πολιτικό αδιέξοδο θα χρειαστεί να διατυπώσουμε γλώσσα ενθαρρυντική σε σχέση με την πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την πορεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις σχέσεις με τους γείτονες. Ευχαριστώ. ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Χάουιτ για το έργο του και για την έκθεση που μας ε, ενημερώνει πάρα πολύ για θέματα για τη Μακεδονία. Υποστηρίζω τις προτάσεις του εισηγητή για αναβολή της ψηφοφορίας. Γιατί η Ελλάδα ως τώρα ήταν η μοναδική χώρα που μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις. Οι Μακεδονές πολιτικοί όμως το φαίνεται ότι και αυτοί έχουν την δυνατότητα και μάλλον θα ενδεχομένως να παρεμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναξη των διαπραγματεύσεων. Αν υπάρχει οποιαδήποτε κίνδυνος να μην υπάρξει αυτό, αυτό ε, θα ήταν πρόβλημα. Ακόμα και αν η Ελλάδα ε, έπρεπε σοφά και έλεγε τώρα αμέσως να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και πάλι θα είχαμε λόγους να περιμένουμε στην παρούσα φάση μέχρι ότου να ρυθμίσουν τα του οίκου τους. Ο εισηγητής ε, αναφέρθηκε σε κάποιες από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Να μιλήσω για δύο εξ αυτών. Για την επτά. αναφέρει ότι το θέμα του ονόματος θα πρέπει να επιληθεί προς το τέλος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης πριν την ε, προσχώρηση. Αναφέρεται μια προφορική τροπολογία. Θα θέλαμε να ακούσουμε ποια είναι αυτή η τροπολογία. Δεν θέλω να την απορρίψω χωρίς να την ακούσω. Αλλά μπορεί να πρόκειται για μια πραγματική διάσταση απόψεων. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επιληθεί το θέμα πριν την ένταξη, αλλά ότι πρόκειται για κάτι εντελώ διαφορετικό από την διαδικασία της προσχώρησης, που θα πρέπει να έχει να λαμβάνει υπόψη μόνο τα σχετικά κριτήρια. Γιατί το να αναφέρουμε ότι το θέμα του ονόματος θα πρέπει να επιληθεί πριν την αρχή των διαπραγματεύσεων, τα μπλέκει. Μπλέκει το θέμα με την, ε, του ονόματος με το θέμα των διαπραγματεύσεων. Στην 53 αναφέρεστε στην διαδικασία ελέγχου που δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν την έγκριση του Συμβουλίου. Το αναγνωρίζουμε αυτό και γι' αυτό προχωρούμε σε προσεκτική διατύπωση. Ζητάμε από το Συμβούλιο να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει αυτή η επιτήρηση, αυτός ο έλεγχος δείχνοντας ε, τη δέσμευση των μεταρρυθμίσεων στην Μακεδονία, ακόμα και αν ε, υπάρχει μπλοκάρισμα πλευράς Ελλάδας για άλλους λόγους. Ε, μπορούμε λοιπόν να το εξετάσουμε αυτό, προκειμένου να συνάδει με τις συνθήκες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για τις τελευταίες τα τελευταία ενημερωτικά στοιχεία που μας έδωσε για την κατάσταση στη Φύρο. Πράγματι μας ανησυχεί όλους η κατάσταση που υπάρχει, η πολιτική κρίση που δεν έχει ξεπεραστεί και από αυτή την άποψη, έχοντας και την εμπειρία ως εισηγητής της έκθεσης για την Αλβανία, σωστά και τότε, όσο υπήρχε πολιτική κρίση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε ουσιαστική δουλειά. Με αυτή την έννοια ε, συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή για την αναβολή της ψηφοφορίας. Θέλω όμως σε σχέση με την πολιτική κρίση να κάνω κάποιες ε, σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτο, όσο υπάρχει η πολιτική κρίση που εύχομαι να λήξει το συντομότερο δυνατό, δεν μπορούν να συζητηθούν προφανώς ουσιαστικά τα προβλήματα που υπάρχουν, αυτά που υπογραμμίζουμε, ενδεχομένως αυτά που έχουμε διαφορετική γνώμη, διότι ενσωματώνονται μέσα στις αντιπαραθέσεις και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Την κρίση και την πολιτική ομαλοποίηση που εύχομαι να επέλθει το συντομότερο δυνατό, για να μπορούν να συζητηθούν τα ουσιαστικά ζητήματα, θα την επιφέρουν, θα την επιλέξουν. Είναι ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων του κράτους, της ΦΥΡΟ. Αυτοί θα το λύσουν το πρόβλημα. Και τρίτο, επειδή η πολιτική κρίση, όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία και από την παρακολούθηση της κατάστασης, είναι, έχει στο υπέδαφος της έντονα φαινόμενα οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, θα έλεγα, μπαίνοντα στην έκθεση, αναφερόμενος σε μία τροπολογία που έχουμε καταθέσει, ότι τα στοιχεία της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης είναι πιο έντονα από αυτά που δίνει η έκθεση. Αναφέρομαι μόνο στο θέμα της ανεργίας των νέων ως χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σχεδόν πλησιάζει το 60% και η τροπολογία έχει το χαρακτήρα και στον εισηγητή μας και σε όλους μας να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι επισημάνσεις μπορούν να γίνουν. Αν δεν δίδεται η πραγματική εικόνα, αν δεν δίδεται ένα κίνητρο να αντιμετωπιστούν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, εν τέλει, λέω και σε τελική ανάλυση, δεν, δεν θα αντιμετωπιστεί και η πολιτική κρίση. Τώρα, δύο-τρει παρατηρήσει με βάση και τι τροπολογίε που έχουμε καταθέσει ε, σχετικά με το κείμενο και με τη συζήτηση που κάθε φορά που συζητάμε την έκθεση τη ΦΥΡΟΜ γίνεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι λαθεμένος ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ένταξης της ΦΥΡΟΜ ως ένα πρόβλημα που τον μπλοκάρει η Ελλάδα. Είναι λάθος. Δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η παρανόηση. Σας το λέει κάποιος που δεν ανήκει σε κυβερνητικό κόμμα, που δεν είμαστε κυβέρνηση στην Ελλάδα για να υπερασπιστώ την κυβερνητική στάση τη σημερινή ή τη χθεσινή. Είμαστε στην αντιπολίτευση δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα λέγοντας ότι η Ελλάδα τον μπλοκάρει και όταν το ξεμπλοκάρει η Ελλάδα όλα θα πάνε καλά. Με αυτή την έννοια οι παρατηρήσεις όσο αφορά το κείμενο γνωρίζω τις διαφωνίες. Ε, τις γνωρίζει βεβαίως και ο εισηγητής, είναι γνωστές. Έχουν να κάνουν πρώτο. κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να ζητάμε να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες και μετά να αντιμετωπιστεί το θέμα του προβλήματος. Είναι σαν να ξεπερνάμε μια διαδικασία χρονοβόρα, επίπονη, με πολλά προβλήματα επίλυσης του θέματος μέσα στο πλαίσιο του ΕΕ, ΟΗΕ. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία, δεν μπορεί να γίνει με άλλον τρόπο. Αν εισηγούμεθα μια διαφορετική σειρά των πραγμάτων, φοβάμαι ότι δεν βοηθάμε, μπορεί να μην συμφωνώ εγώ ή και κάποιοι άλλοι, αλλά δεν βοηθάμε και στην αντιμετώπιση των εσωτερικών προβλημάτων στη γειτονική από τη χώρα μου χώρα. Δεύτερο, νομίζω και δεν βοηθάμε και γι' αυτό έχω καταθέσει και σχετική τροπολογία και δεν νομίζω ότι ο εισηγητής εκεί αποδίδει σωστά τα πράγματα όταν λέει ότι ο όρος μακεδονικός μακεδονική χρησιμοποιείται κατά κανόνα από τον ΟΗΕ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η απόφαση του ΟΗΕ είναι ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι προσωρινοί μέχρι την εξέβρεση της λύσης με βάση τη διαδικασία που έχει κινηθεί. Αν λοιπόν θέτουμε αυτό ότι είναι ο κανόνας, είναι σαν να προδικάζουμε κατά τη γνώμη μου τη λύση της ονομασίας και να δημιουργούμε περαιτέρω δυσκολίες. Αυτή είναι η δική μου η πρόταση. Αυτές είναι οι βασικές παρατηρήσεις συν ε, τη γενική παρατήρηση που έχει σχέση και με την πρώτη εκτίμηση που έκανα. Αν έχουμε την εντύπωση ότι το θέμα της ονομασίας είναι ένα διμερές πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Φύρων, αν το θέμα αυτό το βάζουμε ως σε μια ξεχωριστή παράγραφος και όχι στο θέμα σχέσεων καλής γειτονίας που σημαίνει ότι είναι ένα γενικότερο διεθνές πρόβλημα και πρέπει να λυθεί με αυτές τις διαδικασίες, κατά τη γνώμη μου δεν βοηθούμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος και εύχομαι να το ξαναδεί ο εισηγητής μας. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, αλλά τουλάχιστον ας το ξανασκεφτεί όσο αφορά το που θέτει αυτό το θέμα, γιατί έχει και τη συμβολική του σημασία. Τελειώνω με μόνο την υπενθύμηση ότι παρατηρήσεις που έχουν σχέση με την οικονομική κατάσταση και τροπολογίες ε, νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έχω καταθέσει σχετική τροπολογία, δεν θέλω να φάω περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Oh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Χάουιτ, το οποίο μας παρουσίασε μια, θα έλεγα, ισορροπημένη έκθεση. Ε, εγώ υποστηρίζω κάποιες από τις τροπολογίες των συναδέλφων, όπως την 31, είναι μια βασική αρχή για τις διμερείς σχέσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να εμποδίζουν μια χώρα να προοδεύσει εφόσον θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει ό,τι χρειάζεται γι' αυτό. Ε, επίσης την τροπολογία 40 ε, για την λεγόμενη αρχή της ρεγκάτα όπως λέγαμε δηλαδή ότι κάθε χώρα θα πρέπει να κρίνεται ατομικά και όχι σε σχέση με τις περιφερειακές εξελίξεις ε, τις τροπολογίες που ζητούν από την αντιπολίτευση να επιστρέψει στην Εθνοσυνέλευση ή το, Κοινοβούλιο είναι ο χώρος όπου θα γίνει η πολιτική αντιπαράθεση, η αντιπαράθεση και η μαζική παρέτηση από το Κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο δεν έχει νόημα. Υποστηρίζω την 121 για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δικαστικό και την 129 νομίζω της κυρίας Μακοβέη για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, σαν εισηγητή για το Μαυροβούνιο να πω ότι το Μαυροβούνιο δεν ήταν υποψήφια χώρα κάποτε και διαπραγματεύεται ε, σήμερα με μας. Ε, η Μακεδονία λέει ο μιλητής ήταν υποψήφια εδώ και πάρα πολύ καιρό και βρίσκεται πολύ πιο πίσω πάλι και από ό,τι φαίνεται και το θέμα του ονόματος καθυστερεί τη συγκεκριμένη χώρα θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε να υπάρξει μια λύση. Ας ελπίσουμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η κρίση αυτή σε επίπεδο αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας να επιληθεί, να βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ νέου να κάνει μια θετική σύσταση προς το Συμβούλιο που θα διευκολύνει την διαδικασία ένταξης της χώρας. Κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, αντίστοιχη συζήτηση έχουμε κάνει επαλληλειμμένως, κάθε χρόνο δηλαδή για την ε, πρώην Κουσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αλλά το ερώτημα είναι σήμερα, ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της χώρας αυτής. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα εμποδίζει την ένταξή της. Όχι, η ίδια η έκθεση περιγράφει τα πραγματικά προβλήματα δηλαδή την ανεπάρκεια στο δικαστικό σύστημα, τη διαφθορά, την μη πλήρη εφαρμογή των ελευθεριών των δημοσιογράφων και του τύπου ακόμα και βεβαίως παραλείπει η έκθεση να σημειώσει ότι η διαδικασία που συνεχίζεται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το θέμα του ονόματος που δεν είναι διμερές πρόβλημα αλλά διεθνές βρίσκει αντίθετη την ίδια τη δημοκρατία αυτή. Στην τελευταία συνάντηση του κυρίου Νίμιτς έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις από την Ελλάδα και δεν υπήρξε καν απάντηση από την άλλη πλευρά. Επομένως ε, είναι, επιτρέψτε μου να πω κύριε συνάδελφε, αρκετά υποκριτική η θεωρία ότι στη χώρα αυτή όλα πηγαίνουν θαυμάσια, πρέπει να γίνει μέλος της Ένωσης, αλλά η Ελλάδα την εμποδίζει να ενταχθεί. Και αυτό το αποδεικνύει πολύ περισσότερο η πρόταση που γίνεται για να αναβληθεί η ψήφιση. Η χώρα πέραν των άλλων προβλημάτων έχει ένα ανεπαρκές και αδύναμο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν λειτουργεί. Η αντιπολίτευση δεν είναι στη Βουλή. Αυτό αποτελεί λόγο να αναβάλουμε την ψηφοφορία γιατί νομίζουμε ότι όλα θα έχουν τακτοποιηθεί μέχρι τότε και θα μπορούμε πριν από τον Ιούνιο να κάνουμε μια ωραία έκθεση όπου όλα θα περιγράφονται σωστά. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι πολιτική στάση αυτή. Είναι εκτός πραγματικότητος. Και συνιστώ στην Επιτροπή να προχωρήσει τη διαδικασία ψήφισης στην οποία να αποτυπώνεται η πραγματικότητα. Γιατί πρέπει να αποκριβεί η πραγματικότητα και να αναβληθεί η ψηφοφορία. Αυτό είναι πολιτική στάση. Θεωρώ ότι είναι... Δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω τη στάση αυτή, αλλά δεν είναι πολιτική στάση. Η έκθεση πρέπει να αποτυπώνει την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Και η πραγματικότητα είναι δεδομένη. Πίσω από τις γραμμές της έκθεσης που θέλει να συγκαλύψει την πραγματικότητα, φαίνονται τα γεγονότα. Επομένως δεν βρίσκω κανένα λόγο αναβολής αυτής της έκθεσης με την ελπίδα ότι τα πράγματα θα έχουν δηλαδή τύπης αποκατασταθεί. Η κατάσταση στη χώρα αυτή δεν μπορεί να εξομαλυνθεί. Και αν δεν το καταλαβαίνει η Επιτροπή, καλό είναι άνθρωποι αντικειμενικοί να πάνε επιτόπου για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Γιατί δεν είναι μόνο οι βαθιές αντιθέσεις, αλλά είναι η πολιτική που ασκείται εκεί από όσου έχουν την ισχύ στη δεδομένη στιγμή που οξύνει τις αντιθέσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δημιουργώντας σχέσεις κακής γειτονίας. Και πάντως δεν μπορούν να υπάρχουν διπλά στάνταρ, δηλαδή άλλοι να πρέπει να λύσουν τα προβλήματα για να μπουν στην Ένωση και άλλοι να πρέπει να μπουν στην Ένωση για να μην τα λύσουν ποτέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <coughs> Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιστρέψτε μου και εμένα να συγχαρώ τον ε, κύριο Χαουή, τον εισηγητή, για τη δύσκολη δουλειά που έχει λάβει, Τα μεγάλα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει και την ενεργητικότητα που δείχνει στην προσπάθεια για τη χώρα αυτή. Αναμφίβολα όλοι ενδιαφερόμεθα για την διαδικασία προσχώρησης μιας χώρας σε μια τόσο σημαντική άλλωστε περιοχή. Για τα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί θα αποτελεί και την υποθήκη για τη σταθερότητα στο μέλλον. Για την πρόταση τώρα για την αναβολή θα τοποθετηθώ αμέσως λέγοντας ότι είναι όντως πολύ ασταθής η κατάσταση, πολύ αβέβαιη και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο και να περιμένουμε. Αλλά επιτρέψτε μου να επισημάνω και το εξή με απόλυτη ειλικρίνεια, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είχαν ε, γίνει αντιληπτά στη χώρα αυτή για κάποιο διάστημα και ίσως το θέμα αυτό με το όνομα, ίσως κάποιοι που είχαν έτσι μια καλό, καλή διάθεση, θέλαν να πούν ότι τα πάντα είναι καλά. Ε, τώρα αυτά τα πράγματα βγαίνουν στη φόρα. Εγώ είχα πολλές ανησυχίες και επιφυλάξεις προς τις δημοκρατικές προδιαγραφές για τις σχέσεις με όλους εκείνους που ε, θεωρούν ή ε, αυτοπεριγράφοντας προερχόμενα από μια διαφορετική εθνοτική ε, ομάδα, οικονομικά ζητήματα κτλ. Όλα αυτά λοιπόν κάπως είχαν λησμονηθεί. Ίσως κάποιοι από τους συναδέλφους να μην γνωρίζουν ε, τις λεπτομέρειες αυτών των περιστατικών του Δεκεμβρίου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συζητηθούν γιατί είναι πολύ σημαντικά και στην Ευρώπη αλλά και, και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εάν δει κανεί να μπαίνει αστυνομία μέσα στο κοινοβούλιο και να πετάει έξω από την πόρτα βουλευτή τη αντιπολίτευσης βουλευτές συγκεκριμένα της αντιπολίτευσης. Σημειώνω δε ότι είχε προηγηθεί αντίστοιχη ε, ε, εκδίωξη των δημοσιογράφων από το κτίριο της Βουλής προκειμένου να μπορούν να παρακολουθήσουν την κατάσταση. Άρα λοιπόν εκεί θα ανησυχούσαμε όπου και να συνέβαινε. Λοιπόν, δεν έκανε μόνο ο Καλ Μπίλτ δηλώσεις για την ε, κατάσταση και τα περιστατικά αυτά και η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει και όταν είμαστε επικριτικοί για την ε, έναντι τη αντιπολίτευση για το ότι δεν επανέρχεται στι συνομιλίε, στις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο κτλ. Και συμφωνώ σε αυτό, θα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη στάση. Αλλά για να σα πω, όταν κάποιον, κάποιον τον έχουν πετάξει έξω από το Κοινοβούλιο, πώ θα ζητήσουμε από το κόμμα του να γυρίσει σε μια διαδικασία συνομιλιών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τηρήσουμε ίσες αποστάσεις και να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα για το φαινόμενο αυτό της εκδίωξης από το ε, κοινοβούλιο της αστυνομίας. Και σας ερωτώ, θα τολμούσε κάποιο αστυνομικό όργανο χωρίς εντολές ή έστω προστασία άνωθεν να προβεί σε μια τέτοια πράξη. Λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε επικοδομητική στάση πρέπει να τα πούμε όλα Ιδάλλως αποδυναμώνεται η δημοκρατία και δεν νομίζω ότι θα φέρουμε αποτελέσματα θετικά. Πρέπει και πιέσει να ασκήσουμε και να πούμε τι πιστεύουμε για τις δημοκρατικές προδιαγραφές και τα πρότυπα στη χώρα αυτή και κυρίως της συγκεκριμένη κυβερνήσεως, η οποία κατά με δεν έχει επιδείξει δημοκρατική αξιοπιστία. Και αυτό εξ αρχή, αλλά εμείς προσφύγουμε να δεν το παρατηρούμε. Ο κύριος Πόσιλτ. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι έχουμε να κάνουμε μια έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο του έτους 2011 ε, κατά τη διάρκεια της οποίας η Μακεδονία, και το επαναλαμβάνω, Μακεδονία, Μακεδονία, Μακεδονία, Μακεδονία, Μακεδονία, έχει παρουσιάσει καταπληκτική πρόοδο. Πρόκειται για μια έκθεση πρόοδου, η οποία φυσικά δεν παραγνωρίζει τα ε, κρίσιμα σημεία, τα σημεία επίκρισης. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε εκείνη η χρονιά τι είδους χαρακτηριστικά παρουσιάζει για την πρόοδο της χώρας αυτής. Και ο κύριος Χάουιτ έχει κατά την άποψή μου καταγράψει, ε, καταρτήσει ένα καταπληκτικό έγγραφο, πάρα πολύ σωστά σταθμισμένο και ισορροπημένο και συμφωνώ απολύτως και συμμερίζομαι και υποστηρίζω πλήρως την προσέγγιση του ότι δεν θα πρέπει οι εσωτερικές εδώ αντιπαραθέσεις που διεξάγονται μέσα στο κοινοβούλιο να παρακολουθούν τις αντιπαραθέσεις μέσα στη χώρα. Γιατί πρέπει να δείξουμε στα ε, κόμματα της Μακεδονίας ότι έχουμε μια κοινή ενιαία γραμμή που είναι τήρηση των κριτηρίων για την ένταξη και αυτό να το πούμε για τα κόμματα της Μακεδονίας ώστε να καταλάβουν ότι είναι σαφώς ανοιχτός ο δρόμος για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μαζί τους θα συνεργαστούμε, ότι δεν θα συμπεριφερθούμε κατά τρόπο ανεύθυνο, ότι δεν θα περιπέσουμε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις μαζί τους, ότι τους κάνουμε κακό, δεν θα παραβλάψουμε τη διαδικασία της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει σαφώς συνένεση μεταξύ των κύριων δυνάμεων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι πεπισμένος ότι ο συνέλφος κύριος Χάουιτ έχει καταγράψει τη συνένεση αυτή ξεκάθαρα και με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Η δε πρόταση για αναβολή ενδεχομένως να φαίνεται λογική. Την υποστηρίζω και εγώ, αλλά αντιλαμβάνομαι και την δυσφορία του συναδέλφου Χάουιτ και τη δυσκολία που έχει στο να αποδεχθεί την πρόταση αυτή. Αυτό το αισθάνομαι και εγώ ακόμη περισσότερο ε, έχοντας ακούσει το δεύτερο κομμάτι της συζητήσεως, διότι υφίσταται ο κίνδυνος αυτή η αρχή, εκ πρώτης όψεως ε, λογική ε, αναβολή είτε να παρερμηνευθεί είτε να τύχει καταχρήσεων, να πέσει θέμα καταχρήσεων. Και υπογραμμίζω δεν πρέπει ούτε να παρερμηνευτεί ούτε να πέσει θέμα καταχρήσεων. Πρώτον για από εκείνου που ε, στη χώρα είτε προκαλούν είτε μποϊκοτάρουν ώστε να ενθαρρυνθούν και στην περαιτέρω στη συνέχιση των προκλήσεων και της αποχής γιατί δεν αναβάλουμε την ψηφοφορία προκειμένου να τους ενισχύσουμε και να ε, ενδυναμώσουμε τη θέση τους και τις δυσκολίες που θέτουν στην συζήτηση. Αντιθέτως, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε σε μια συνενετική λύση. Σημείο 2. Δεν αποτελεί αυτή η αναβολή ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο ώστε για αναβολή των διαπραγματεύσεων. Η κυρία Γιαννάκου μιλάει για ένταξη. Μα δεν μιλούμε, δεν βρισκόμαστε ενώπιον εντάξεως. Δέκα χρόνια πέρασαν για να αναγνωριστεί το καθεστώς υποψηφίου κράτους, δέκα χρόνια για την αναγνώριση του καθεστώτος ε, υποψηφίου κράτους, ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Περί αυτού πρόκειται. Η αναβολή λοιπόν για μερικές εβδομάδες ε, της ψηφοφορίας δεν θα πρέπει να πέσει θύμα της καταχρήσεως εκείνων που δεν θέλουν να επιτρέψουν ε, τις διαπραγματεύσεις και θέλουν να τις καθυστερήσουν. Και επιπλέον δεν θα πρέπει η αναβολή αυτή των της εκθέσεως, της ψηφοφορίας εκθέσεως, δεν θα πρέπει να πέσει θύμα των καταχρέσεων ε, και, αναβολή, και να οδηγήσει σε αναβολή των διαπραγματεύσεων ούτε πρέπει να πέσει θύμα της ε, καταχρήσεως του ε, λεγόμενου εκείνου ονόματος, του ζητήματος του ονόματος. Το λέω λεγόμενο διότι δεν υπάρχει ζήτημα ονόματος, ούτε ευρωπαϊκό, ούτε δε, ε, διμερές, ούτε διεθνές πρόβλημα υπάρχει. Πέραν της Ελλάδος δεν υπάρχει κράτος το οποίο να έχει θέσει ζήτημα ονόματος. Πρόβλημα υπάρχει μόνο στο μυαλό ορισμένων Ελλήνων πολιτικών, λέει ο μιλητή. Και είμαι πεπισμένο απολύτω ότι πια πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία και πρέπει να αλλάξει η ονομασία του κράτους. Υπάρχουν συμφωνίες, ήδη υπάρχει μια συνένεση ευρύτερη σε αυτό. Πρέπει λοιπόν να αναγνωριστεί ότι η Μακεδονία πρέπει να ονομάζεται Μακεδονία με το ίδιο δικαίωμα που και εμείς ονομαζόμαστε Βαβαρία. Είναι παράλογο να συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι, λέει ο μιλητή. Γι' αυτό λοιπόν λέω ναι ξεκάθαρα για την πρόταση του κυρίου Χάουιτ, του Χάουιτ, αλλά να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε η αδίποτε προσπάθεια είτε ε, κατάχρηση αυτών, η εκμετάλλευση αυτή τη αναβολή. Ο κύριος Κατσίν. Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεται. Το μικρόφωνο του κυρίου Κατσίνη είναι αναμένο αλλά δεν ακούγεται τίποτα. Ο σκιώτη μα, ο κύριο Νικολάτσιν, δεν είναι εδώ σήμερα δυστυχώ. Αλλά να ε, διαβιβάσω το μήνυμά τη, να σα συγχαρώ για τη δουλειά σα, για την ισορροπημένη σα έκθεση, για τον ενθουσιασμό και τη θετική ενέργεια που δαπανίσατε στο θέμα της Μακεδονίας, στις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Μακεδονία και για να δημιουργηθεί μια πολύ καλύτερη ατμόσφαιρα. Από την άλλη να πω ότι ο υψηλός, υψηλού επίπεδου πολιτικός διάλογος δεν μπορεί να αντικαταθιστήσει τη διαδικασία α, ένταξης. Αυτό αναζητούμε. Δυστυχώς οι πρόσφατες εξελίξεις δημιούργησαν μια νέα κατάσταση. Η έκθεσή σας αποτυπώνει με θετικό τρόπο και σας υποστηρίζουμε, αλλά καθίσταται η έκθεσή σας αυτή εικονική, όλο και πιο εικονική, γιατί η πραγματικότητα είναι διαφορετική και αρνητική και η πραγματικότητα απέχει πολύ από την έκθεση που την πραγματικότητα της έκθεσή σας. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η αναβολή είναι ένας καλός εμβιβασμός. Και φυσικά πάντα θα υπάρχει το θέμα και μια μάχη για το, την ερμηνεία της αναβολής αυτής. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που ήθελα να αναφέρω. Ο Στέφανος Στανίνου ήταν εκεί, μετέβη εκεί πολλές φορές και ο, Επίτροπες, Επίτροπος προσπάθησε να δημιουργήσει τους όρους για να κάνει, να αποστείλει ένα θετικό μήνυμα και τελικά αναγκάστηκε να αναβάλει την επίσκεψή του. Γιατί η Μακεδονία βυθίζεται, βυθίζεται σε ένα πολιτικό α, χάος. Και θα ήθελα να καλέσουμε την ευκαιρία αυτή της πολιτικές ελίτ της Μακεδονίας να κοιταχτούν στον καθρέφτη με ρεαλιστικό τρόπο και να σταματήσουν να κατηγορούν οι μεν τους δε. Θα πρέπει να βρεθεί μία λύση. Να, να, να θυμίσω και κάτι άλλο από τη, τα Βαλκάνη ή ο Πρωθυπουργό της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου ε, συνέρχονται σε κάθε περίπτωση που μπορούν. Την, για έκτη φορά θα ε, συνέλθουν εδώ στις Βρυξέλλες στις 4 Μαρτίου. Αυτό είναι διάλογος υψηλού επίπεδου. Δεν έχουν όμως μεταξύ τους επικοινωνία. Είναι μια στιγμή αλήθειας. Και θα πρέπει να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα και τώρα να μιλήσω τη δική μου γλώσσα, γιατί θέλω κάτι να πω για την εθνική ταυτότητα και θα θέλω να μιλήσω σε σλάβικη γλώσσα. Εγώ είμαι από την Σλοβενία και μιλώ την σλοβενική γλώσσα, η οποία συγκαταλέγεται στις ε, σλαβικές ε, γλώσσες. Και αυτό γινόταν στα Δυτικά Βαλκάνια πριν από κάποιο καιρό. Υπάρχουν δύο σλαβικά έθνη, τους Βούλγαρους και τους Μακεδόνες. Έχουν τους ίδιους Αγίους, έχουν τους ίδιους ποιητές, επισκέπτονται τα ίδια μοναστήρια. Και τώρα ακούμε ότι οι Μακεδόνες δεν είναι πλέον Σλαβοί. Μιλούν σλαβική γλώσσα χρησιμοποιούν το κυριλικό αλφάβητο, χρησιμοποιούν την ίδια γραμματική, αλλά δεν είναι Σλάβοι πια. Και οι Βούλγαροι λοιπόν. Η πολιτική ελίτ στη Μακεδονία θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι προκαλεί μεγάλη ζημιά και στις σχέσεις με τους γειτονές της. Αν και άλλοι άλλα έθνη σλαβικής καταγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια αρχίσουν με τον ίδιο τρόπο να ξαναγράφουν την ιστορία τους, θα καταλήξουμε τελικά σε έναν εκβαλκανισμό όλη τη Ευρώπη, τη Ευρώπη με το χείριστο τρόπο. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση θα πρέπει να καλέσουμε και τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού και την αντιπολίτευση να επιστρέψουν από την προϊστορία στη σημερινή εποχή και να μας επιτρέψουν εδώ στο Κοινοβούλιο να εγκρίνουμε την έκθεση για την έκθεση προ του 2012. Αλλά θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα προς τα εμπρός και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Και μόνο τότε θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τον εισηγητή και να βοηθήσουμε και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν υπόψη τη σύσταση και να προβλέψουν μια ημερομηνία για την Μακεδονία. Ξέρω ότι τα λόγια μου ακούγονται στη Μακεδονία και ξέρω ότι αυτό θα αποτελέσει μια τεράστια πρόκληση στον εισηγητή, για τον εισηγητή που κάθεται εδώ στην αίθουσα. Θα είναι και μια μεγάλη πρόκληση για εκείνους που θα πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσο θα δημοσιεύσουν αυτά ή όχι. Αλλά μόνο η ίδια η Μακεδονία μπορεί να βοηθήσει και τον ίδιο στον εαυτό και την ε, Βουλγαρία και άλλες χώρες για μια θετικό αντίκτυπο και μια ημερομηνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σκούκαν. Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Κουμουτσάκος. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πολιτική κατάσταση στα Σκόπια είναι πολύ προβληματική. Οι θεσμοί ίσα ίσα που λειτουργούν, τα δημοκρατικά πρότυπα καταπατώνται καθημερινά και στο σύνολό της ε, η δημοκρατία πάσχει. Παρά την ε, κατάσταση είπατε ότι δεν θα πρέπει να τους αποθαρρύνουμε και να τους εξαπατούμε. Και βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με μια λίγο περίεργη κατάσταση. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και ομαλά στην πρώην δημοκρατική στην δημοκρατία της Μακεδονίας, μας λέτε ότι θα πρέπει να αποστέλουμε θετικά μηνύματα και να τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν. Όταν τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, λέμε και πάλι ότι δεν θα πρέπει να τους αποθαρρύνουμε. Έμα, ε, ας αποφασίσουμε. Είτε όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά θα τους ενθαρρύνουμε και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά θα τους αποθαρρύνουμε, θα τους ασκούμε κριτική. Και με επικοδομητικό μάλιστα τρόπο. Δεν είναι δυνατόν πάντα φετικά μηνύματα να αποστέλνουμε ό,τι και να συμβαίνει στη χώρα αυτή. Και μετά να κάνω ένα άλλο σχόλιο. Πάλι κάποιοι συνάδελφοι έθεσαν στο στόχαστρο την Ελλάδα. Ερωτώ, συνάδελφοι. Ποιος πήρε το λόγο στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να πει ότι δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν ακόμα οι διαπραγματεύσεις. Μόνο η Ελλάδα, όχι, και η Βουλγαρία. Και κάποιες άλλες χώρες, θα έλεγα, ότι έδειξαν κάποια διστακτικότητα ήταν η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Και ξέρετε και τι προβλήματα έχει η Ρουμανία σε ό,τι αφορά την ιστορική κατάσταση που επικρατεί στην ε, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Τι σημαίνει αυτό, ότι τρει όμορε χώρε έχουν σοβαρά προβλήματα με τη χώρα αυτή. Εδώ στο κοινοβούλιο αυτό, στο δημοκρατικό αυτό κοινοβούλιο, δακτυλοδεικνύουμε δύο εταίρους, την Βουλγαρία και την Ελλάδα, και την Αλβανία και λέμε ότι α, αυτές είναι χαζές και ο μοναδικός έξυπνος είναι κ. Κρουέσκι. Τελευταίο σημείο. Όταν κύριε Κούκαν καλείτε τους Μακεδόνες πολιτικούς να κάνουν το χύψη, σκεφτήκατε ποτέ ότι διακινδυνεύετε να λάβετε επιστολές από από τους ε, Μακεδόνες πολιτικούς ε, στην ε, χώρα μου, στην Ελλάδα. Δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες επιστολές, γιατί 30-40 μέλη της Ελληνικής Βουλής εκπροσωπούν τη Μακεδονία της χώρας μου. Γι' αυτή χρησιμοποιείται τον όρο «μακεδονικός» στο κείμενο. Είναι περίπλοκη η κατάσταση, συνάδελφοι, και δύσκολη να προσχωρήσει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον όρο ότι θα επιληθούν όλα τα προβλήματα. Αυτά είχα να πω για να προσθέσω τώρα κάτι στα σοφά λόγια της κυρίας Μαριέτα Γιαννάκου. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πλένκοβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Κουκάνα. Και καταρχάς Θα ήθελα να κάνω πολύ θετικά σχόλια για το έργο του κύριου Χάουιτ, του εισηγητού, τον οποίο πριν από 1,5 χρόνο με διαφορετικό τίτλο συνάντησα στα Σκόπια σε μια διάσκεψη για, και όπου μπόρεσα να δω πόσο αποτελεσματικά προσπαθεί να φέρει την, την Μακεδονία πιο κοντά, τα Σκόπια πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχω μια εμπειρία αντίστοιχη με αυτή της Μακεδονίας να παρουσιάσω πλευρά της Κροατίας για τα τελευταία 15 χρόνια. Το Νοέμβριο του 2000 υπέγραψε στο Ζάγκρεπ την ε, συμφωνία SAA η Μακεδονία. Ε, μια συμφωνία που αποτέλεσε για μας ε, την απαρχή μιας προσπάθειας να ξεφύγουμε από τις πολιτικές, πολιτικώς ορθώς, ορθές προτάσεις και να κάνουμε ουσιαστική δουλειά για την ένταξη που είναι μπροστά μας τώρα πια. Η Μακεδονία είναι υποψήφια χώρα από το 2005. Έχουν ε, αρχίσει από το 2009 να απευθύνονται κλείσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, Επιτροπή για την Άνοιξη των Διαπραγματεύσεων. Ε, βρίσκεται λοιπόν η χώρα μπροστά σε ένα σενάριο το οποίο μπορεί να προκαλεί και δυστημία και δυσφορία και αίσθημα ματέωσης. Άρα ίσως να είναι ευνόη, να είναι κατανοητές κάποιες καθυστερήσεις στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων πλευράς της χώρας. Ε, πρέπει να την ενθαρρύνουμε λοιπόν, γιατί τα μέσα αυτά της, ε, τα, ε, της υποστήριξης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκολύνουν ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη και η έκθεση αυτή της πρόοδου, η έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καταγράφει πιστεύω πολύ πιστά τα πορίσματα από τον Οκτώβριο του 2012, πρέπει να χαράξει τον δρόμο προς τα μπρος, πρέπει να επανέλθει πιστεύουμε η αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο δεν μπορεί να απέχει από τις εργασίες της Βουλής, δεν είναι ο τρόπος αυτός να λυθούν τα προβλήματα και επίσης με κάθε σεβασμό προς τους Έλληνες φίλους για την επίλυση των προβλημάτων εμείς οι Κροάτες θεωρούμε ότι ο εξευρωπαϊσμός διμερών θεμάτων είναι σφαλμένος τρόπος, δεν είναι ενθαρρυντικός ε, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε άλλωστε μπορεί να βοηθήσει τη διαδικασία της ε, διεύρυνσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you, Miss Ευχαριστώ κυρία Πακ. Συνάδελφοι, αγαπητοί. Κυρία Χάουιτ, να σας συγχαρώ για την έκθεσή σας, πολύ καλή και νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε Θα πρέπει να εξετάσουμε ότι η έκθεση αυτή προόδου δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια για αυτά που συνέβησαν μεταξύ του φθινόπωρου του 2012 και τη σημερινή χρονική στιγμή. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Το ίδιο κάνουμε και με την Βοσνία. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτά που συνέβησαν μέχρι τότε. Το θέμα του ονόματος δεν είναι, όπως είπε η κυρία Γιαννάκου, ένα διεθνές ζήτημα. Όπως είπε ο συνάδελφος Άντρα, είναι ένα διμερές θέμα. Είτε κανείς το καταλαβαίνει, είτε δεν το καταλαβαίνει το θέμα αυτό, είναι αμυγός διμερός. Ούτε η κυρία Πάκου, ούτε ο κύριος Χάουιτ έχει πρόβλημα που η χώρα ονομάζεται Μακεδονία ο συναδέλφος ε, που είπε ότι ο κύριος Κούκαν θα λάβει θυμωμένες επιστολές από τους Μακεδόνες της Ελλάδας. Ε, δεν το καταλαβαίνω. Οι Μακεδόνες που είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι Έλληνες, υποθέτω. Οι Βαβαροί που είναι στο γερμανικό κοινοβούλιο είναι Βαβαροί και Γερμανοί. Οι Μακεδόνες που εκλέχθησαν, ελέγχθησαν ως Έλληνε, όχι ω μακεδόνε, Δεν το καταλαβαίνω. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι το κάνετε εσεί το πρόβλημα. Και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να το αποδεχόμαστε. Το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω. Έφυγε ο συνάδελφο από τη Βουλγαρία βέβαια. Οι τοπικέ εκλογέ που θέλουμε, που πρέπει να θα μποϊκοταριστούν. Έχω ε, εμπειρία στα Βαλκάνια, στην Αλβανία για τις ε, το μποϊκοτάρισμα εκλογών. Σε τοπικές εκλογές, στο Κοινοβούλιο, είναι πολύ μεγάλες οι δυνατότητες μποϊκοταρίσματος. Θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι το μποϊκοτάρισμα δεν είναι δημοκρατικό μέσο. Είναι ανόητο και αφήνει το πεδίο ανοιχτό για τους αντίπαλους φορείς και δείχνει ότι η χώρα δεν είναι όριμη και είμαι σίγουρη ότι η κατάσταση είναι η εξή. Στη Μακεδονία και, τα δύο, και οι δύο πλευρές θέλουν να υπάρξει μελλοντική προσχώρηση στην Ένωση. Υποστηρίζω λοιπόν μία αναβολή της ψηφοφορίας γιατί ελπίζω να διευκολυνθεί η κατάσταση. Κατά δεύτερον, τα προβλήματα στη χώρα αυτή είναι μεγάλα και έχουν διωγγωθεί κι άλλο. Ξέρω ότι όταν έλαβε το 2005 το καθεστώς υποψήφιας χώρας, το είχε πραγματικά κερδίσει με τον υδρότα τη. Αλλά το γεγονό ότι περιμένει ακόμα σήμερα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι πραγματικά παράλογο και έχει να κάνει με τη μία ιστορία αυτή τη συγκεκριμένη, με το όνομα. Το γεγονό ότι στο μεταξύ έχουν διεγκωθεί και άλλα προβλήματα σε σχέση με το 2005 έχει να κάνει με την ε, διαρκή αβεβαιότητα που επικρατεί. Και έτσι όπως και στις γειτονικέ χώρες έχει ε, λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις ο εθνικισμός. Και δεν είμαι βέβαιη. σε σχέση με τα ψέματα της κυβέρνησης ε, σε σχέση με την ιστορία και τους μεγάλους Μακεδόνες. Κοιτάξτε, προκαλεί τους γείτονες. Είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο θα πρέπει να τον διακόψουμε δίνοντας μια ημερομηνία για την προσχώρηση και να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Και να σας πω ότι ε, είναι τεράστια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και θα πρέπει να δώσουμε όμως μια ε, ευκαιρία να ξεχάσετε τα χαζά εθνικιστικά ζητήματα. Θα πρέπει κανείς να έχει την κοινή λογική αυτή. Για να μιλήσω και στους συναδέλφους για την Ελλάδα. Είναι κανείς εδώ από την Ελλάδα? Να σας ρωτήσω. Πώς να αυτό που καλούνται πια αυτοί οι άνθρωποι. Από τον ουρανό έπεσαν. Μακεδόνες είναι αν είστε κι εσείς Μακεδόνες, αν είναι οι ίδιοι Μακεδόνες όπως στην Ελλάδα, αν είναι άλλοι Μακεδόνες ε, που έμεναν σε άλλο τμήμα της Μακεδονίας. Δεν είναι ντροπή. Πώς να αποκαλούνται πρώην Γιουγκοσλάβες. Κάπως πρέπει να έχουν ένα όνομα. και να τους αφήσουμε τουλάχιστον το επίθετο της Μακεδονίας. Δεν μιλάω για ενδεχόμενο όνομα που θα βρεθεί. Γιατί τότε ε, το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καν το επίθετο. Κανείς στην Ελλάδα δεν θέλει να στερηθεί το επίθετο Μακεδόνας, Μακεδονικός, δεν θα πρέπει να το στερούμε λοιπόν και από τους γείτονες. Λίγη αγάπη προς τον πλησίον και θα μπορούσαμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Και η Μακεδονία δεν θα ήταν σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση, η οποία προκλήθηκε εν μέρη και από τα διεθνικά προβλήματα, τα οποία αναπτύχθηκαν λόγω επίσης και της ε, του προβλήματος της ονομασίας. Γιατί για άλλους το, θέμα του ονόματος ε, δεν έχει σημασία, αλλά για άλλους έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ξέρω ότι ε, όσοι είναι εδώ δεν ε, συμφωνούν ότι έχουμε δίκιο, αλλά μόνο οι Έλληνες και οι Βούλγαροι έχουν το πρόβλημα αυτό. Ίσως να υπάρχει μια κρυφή ατζέντα από εκεί πίσω, δεν ξέρω σχετίζεται, αλλά θα ήθελα να τα αφήσουμε αυτά κατά μέρο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μα. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα του δίνω το λόγο στην κυρία Εμπρισάτση και την Προεδρία στον Πρόεδρο. Thank Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δείχνω κατανόηση για ότι ακόμα δεν έχετε ε, μάθει το όνομά μου. Καλύτερα πάντως από ό,τι πριν από δύο μέρες. Άντε, κάνα δύο χρόνια ακόμα και το μάθετε που θα σας πάει. Ο κύριος Πόσελτ χωρίς μικρόφωνο. Και τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα λάβω το λόγο στη μετρική μου γλώσσα. Δεν είναι λοιπόν τόσο εύκολο να παρακολουθούμε αυτά που λέει η Ντόρις. Έκανε πάντως μια πολύ καλή περιγραφή της κατάστασης ε, και συμφωνώ με τα όσα είπε η Ντόρις Πακ. Και ο κύριος Πόσολτς νωρίτερα. Δεν ήθελα να κάνω κάποια σύντομα σχόλια πάντως. Οι συνάδελφοι όσοι τουλάχιστον τάχθηκαν κατά της ε, αναβολής της προφορίας του ψηφίσματος ήταν είτε από τη Βουλγαρία είτε από την Ελλάδα επιτοπλίστων. πλήστον. Είδε Έλληνες στάσου λένε ότι δεν φταίει η Ελλάδα που δεν έχει γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης η Μακεδονία ακόμη Να, αγαπητοί συνάδελφοι, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι θα καταστεί αυτομάτως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Μακεδονία εάν αρθούν οι επιφυλάξεις της Ελλάδας. Αλλά ίσως θα μπορούσε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις εάν δεν παρεμπόδιζε το δρόμο αυτό η Ελλάδα, αν δεν έθετε προσκόμματα. Εδώ ακριβώς είναι όλη η διαφορά. Μεταξύ λοιπόν του αρχίσουν οι διαπραγματεύσει και το να γίνει ένα κράτο μέλο ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και να περάσουν δεκαετίε. Η δική μου η πατρίδα, η Σουηδία, πέρασε πάνω από πέντε χρόνια σε διαπραγματεύσει πριν να γίνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και φαντάζομαι ότι μπορεί κανεί να συγκρίνει την δημοκρατική, οικονομική, πολιτική απόσταση ε, μια Σουηδία που έχει περάσει πάνω από 200 χρόνια χωρί πόλεμο με μια χώρα των Βαλκανίων. Αλλά ακόμα και η Σουηδία μπόρεσε μόνο ύστερα από πέντε χρόνια να ανταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα φανταστείτε πόσε δυσκολίε και χρόνο έχει μπροστά η Μακεδονία για να ολοκληρώσει τι διαπραγματεύσει. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τη Μακεδονία, αλλά για όλε τι χώρε τη Δυτική Βαλκανική, γιατί έχουν πολλή δουλειά μπροστά του. Όμω ο καλύτερο τρόπο για να γίνουν οι σχετικέ μεταρρυθμίσει είναι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Αυτό ακριβώ είναι το επιχείρημα που προβλήθηκε και εν ώψη τη ενάρξη των διαπραγματεύσεων με την Κροατία και για το Μαυροβούνιο επίση ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ακριβώ προβλήθηκε και σε σχέση με τη Σερβία αλλά και με τη Μακεδονία σαν επιχείρημα. Είχαμε επισημάνει ότι χρειάζεται ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Διότι προφανώς με το που αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις έχουμε και την περισσότερη δυνατότητα, τη μεγαλύτερη μόχλευση εμείς να πιέσουμε και να οθήσουμε τα πράγματα προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να βελτιωθούν. Και τώρα αν μου επιτρέπετε θα επιθύνω λίγο το λόγο στους Έλληνες συναδέλφους. Γιώργο, είπες ότι δεν εμποδίζει ή δεν εμπόδισε η Ελλάδα αλλά και η Βουλγαρία, ότι δεν έχει μόνο η Ελλάδα αλλά και η Βουλγαρία πρόβλημα με την ε, Μακεδονία. Εγώ συμφωνώ με την Doris Πακ. Το 2005, πριν από τόσα χρόνια που δόθηκε το καθεστώς του ε, υποψηφίου κράτους στην ε, Μακεδονία, μόνο η Ελλάδα είχε προβάλει αντιρρήσεις και εμείς είχαμε προειδοποιήσει και είχαμε πει ότι εάν δεν προχωρούσαν οι διαδικασίες των μεταρρυθμίσεων, και αυτό ισχύει για όλα τα κράτη της Δυτικής Βαλκανικής, όχι μόνο για τη Μακεδονία, αλλά αν δεν γινόντουσαν μεταρρυθμίσεις, πολιτικές εντάσει θα προχωρούσαν, εθνικισμοί θα εξελίσσονταν και θα και θα ήταν πολύ χειρότερα τα προβλήματα. Ήταν ένα μήνυμα το οποίο απευθύναμε προ πάσα κατεύθυνση και για άλλε χώρε και γι' αυτό άλλωστε καλέσαμε και για την άνοιξη πραγματεύσεων με τη Σερβία, γιατί είναι ο μόνο τρόπο να αντιμετωπίσουμε του εθνικισμού. Ε, το γεγονός ότι δεν έχει μόνο η Ελλάδα πρόβλημα με την ε, Μακεδονία αλλά και η Βουλγαρία για μένα δεν είναι καινοφανές. Το έχουμε ε, επισημάνει εδώ και χρόνια και έχουμε προειδοποιήσει. Όταν άσκησε βέτο στην ένταξη της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα αλλά και στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο πιο πολύ καθυστερεί και δεν θα είναι μόνο η Βουλγαρία και η Ελλάδα κατά της ε, Μακεδονίας αλλά και άλλες βαλκανικές χώρες θα εντείνονται διαρκώς οι εντάσεις και οι εθνικισμοί και θα καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να λάβουν χώρα. Γι' αυτό αγαπητοί φίλοι, όπως και όλες οι άλλες χώρες στη Βαλκανική, ε, Όπω και για όλε τι άλλε χώρε στη Βαλκανική, αν θέλουμε αλλαγέ, αν θέλουμε εξελίξει, αν θέλουμε μεταρρυθμίσει και δημοκρατία, αυτό που χρειαζόμαστε εν τέλει είναι να κάνουμε ακόμη ένα βήμα, να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο και έτσι να μπορέσει κάθε χώρα να αναπτύξει μια ε, προοδευτική διαδικασία για την προσχώρηση. Η Μακεδονία παραμένει ε, στο Προφάλαμο, περιμένει με αδημονία εδώ και χρόνια. Ε, πρέπει κάπως ε, να τους βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να περιμένουν επαόριστον και πρέπει να τους επιτρέψουμε να πραγματοποιήσουν πρόοδο το ταχύτερο δυνατό. Εγώ συγχαίρω τον κύριο Χάουιτ για το εξαίρετο κείμενο του ψηφίσματός του, της προτάσεώς του. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε με τις συνομιτικές προτάσεις να βρούμε την καλύτερη και αποδεκτή για όλους λύση και εύχομαι κάθε δυνατή επιτυχία. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα επανεξετάσετε τις εξελίξεις στη χώρα αυτή τις επόμενες εβδομάδες. Πάντως, οι εκτιμήσεις μας συμπίπτουν με τις εκτιμήσεις που κάνατε και οι περισσότεροι από εσά και με τις οποίες είχαμε κάνει πέρυσι. Όταν τον προηγούμενο χρόνο εκδώσαμε την έκθεση πρόοδου, κυκλοφόρησε η, έκθεση, η έκθεση πρόοδου, είπαμε ότι ο διάλογος υψηλού επίπεδου βοήθησε. Υπογραμμίσαμε επίσης και κάποιες προκλήσεις και κάποιες δυσκολίες οι οποίες υπήρχαν. Πάντως πιστεύουμε ότι μόνο στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων θα μπορέσουμε τις δυσκολίες αυτές να τις αντιμετωπίσουμε πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να περάσουμε στο επόμενο στάδιο για να διασφαλίσουμε την ειρήνη, την ηρεμία και να μην μεγενθύνουμε τους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να παρουσιαστούν. Δεν αμφιβάλλουμε για τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, μας δημιουργεί πρόβλημα η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και η κατάσταση αυτή ακριβώς πιστεύουμε ότι κρατάει ε, πάρα πολύ καιρό και αυτό είναι απαράδεκτο και γι' αυτό ακριβώς οι διεθνείς εταίροι της χώρας όπως και οι Ηνωμένε Πολιτείε ζητούν από τις δύο πλευρές να βρουν μία λύση σύμφωνα με το εθνικό συμφέρον της χώρας. Ζήτησαν επίσης να υπογραμμιστεί η σημασία που έχει η Εθνοσυνέλευση της ΦΥΡΟΜ και ε, η σημασία της σαν εικόνα των δημοκρατικών θεσμών της χώρας. Νομίζω ότι έχουν υπάρξει κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις 24 Δεκεμβρίου και να αποφευθούν τέτοιου είδους συμβάντα στο μέλλον. Μαζί με αρκετές άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ήδη γίνει αντικείμενο α, συζήτησης. Ο Επίτροπος Φιούλε είναι σε επαφή με τις δύο πλευρές, επισκέφθηκε πριν μερικούς μήνες τα Σκόπια ανέβαλε την επίσκεψη που είχε προγραμματίσει την προηγούμενη εβδομάδα για να αξιολογηθεί ο διάλογος υψηλού επίπεδου, θεωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πολιτική συγκυρία δεν προσφέρεται για μια τέτοια συζήτηση και θέλει να δώσει χρόνο στους πολιτικούς ηγέτες της χώρας να βρουν μια λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο διάλογος υψηλού επίπεδου έχει σταματήσει. Εμείς συνεχίζουμε τις επαφές μας σε επίπεδο τεχνικών εμπειρογνωμόνων και προετοιμάζουμε ακριβώς τα πράγματα. Και αυτό ε, μας δημιουργεί, η πολιτική κρίση μας δημιουργεί μια δυσφορία, διότι υπάρχουν στοιχεία στα οποία έχει υπάρξει ε, πρόοδος, έχουν υπάρξει θετικές εξελίξεις. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα συνεχίσουμε τις προπαρασκευαστικές μας προσπάθειες και θα παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Uh, θα πρέπει να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Γιάννη Κασουλίδη που είχα στο τηλέφωνο μόλις τώρα και να σας πω ότι αναλαμβάνει υπουργός των Εξωτερικών. Σας απευθύνει θερμούς χαιρετισμούς. Θα έρθει με την πρώτη ευκαιρία που θα γίνει Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών να σας χαιρετήσει και από κοντά και βέβαια αναλαμβάνει με κάθε αίσθηση ευθύνη σε αυτό το καθήκον του Υπουργείου των Εξωτερικών, των για τη χώρα του σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και θα ήθελα να κάνω μια ε, σύντομη παρατήρηση. Κύριε Χάουιτ, το θέμα της αποχής από τις εργασίες της Βουλής με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όπως υπόθηκε ήδη δεν είναι μία λύση. Το να απέχει κανείς από τις εργασίες της εθνικής αντιπροσωπείας δεν μπορεί να είναι μία υπεύθυνη συμπεριφορά και μόνο κακό μπορεί να κάνει στη χώρα εν όλο. Ξέρουμε ότι το ίδιο ε, έγινε προσπάθεια να αναπτυχθεί σαν δραστηριότητα, η αποχή δηλαδή και στην Αλβανία, κάτι το οποίο όμως ε, ε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά και δεν μπορεί να αποτελέσει για μας λόγο αναβολής. Ε, υπάρχει δηλαδή η προσπάθεια αυτή τη στιγμή να παρεμποδιστεί το, έδρο, το έργο μιας κυβερνήσεως ώστε να καθυστερήσει η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. και εν γέννη βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση η οποία απέχει από τις εργασίες της ε, Βουλής ή μποϊκοτάρει, ε, όπως τουλάχιστον απαιτήθηκε ξεκάθαρα στην Αλβανία, είναι εκείνη που έχει και τα πιο πολλά φτεξίματα. Το ίδιο είδαμε, όπως είπα, στην Αλβανία και, σε σχέση, και βλέπουμε και στη Μακεδονία και σε σχέση με τα μειονοτικά κόμματα. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να μου κάνετε μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα μακεδονικά ε, ή αλβανικά ή το αλβανικό καλύτερα κόμμα, τι είδους ε, πλειοψηφίε εκφράζουν, τι ακριβώς εκφράζουν ε, ως προς τα τμήματα του πληθυσμού. Για το θέμα της ονομασίας πρέπει να σας πω ότι έχει αρχίσει να με κουράζει και να με βαραίνει με βαραίνει εκ μέρους και της, Ευρω... και της ελληνικής πλευράς αλλά και από την άλλη πλευρά με κουράζει. Διότι αν κανείς θέλει και την ε, συνένεση του γείτονα και υποδαβλίζει διαρκώς ε, ένα ζήτημα ονομασίας με το να επικαλείται ε, προέλευση από τον Αλέξανδρο, τότε προφανώς υπάρχει θέμα. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια για ε, δημιουργία, για κατασκευή μιας ταυτότητας που δεν υπήρχε, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με σφετερισμό της ταυτότητας άλλης χώρας. Ε, αυτό προξενεί προφανώς δυσκολίες και είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Ωστόσο, Πρέπει να επισημάνω ότι πρόκειται μόνο για διμερές και όχι για διεθνές ζήτημα. Ένα διμερές ζήτημα το οποίο έχει ως διάμεσολαβητή τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά πρόκειται για διμερές ζήτημα. Ωστόσο θα πρέπει να διερωτηθούμε τι είδους συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τη σταθερότητα όλης της περιοχής. Τι είδους πιέσεις, ε, δυνατότητες δημοσιολάβησης, ανάγκη για συμμετοχή μπορεί να, αποτελέσει, να δημιουργήσει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κοιτάξουμε με πολύ επιφυλακτικό μάτι της, ε, την κατάσταση αυτή. Και πάντως ε, απαραίτητο είναι για μένα να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε να διονύσει αυτή η κατάσταση και θα πρέπει να ασκηθεί ε, ε, πίεση και προς τις δύο πλευρές και σε επίπεδο Συμβουλίου αλλά και, προς τους, και σε επίπεδο μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις δύο πλευρές, επαναλαμβάνω, προς τα δύο κράτη για να προχωρήσουν. γιατί εδώ δεν μπορεί να εξαρτηθεί ούτε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε και το μέλλον το ευρωπαϊκό ενός, ε, μονο, ε, μονομένου κράτους από μόνο το ζήτημα του ονόματος. Ε, δεν έχει συμπεριφερθεί πολύ ευφυώς η χώρα μέχρι τώρα και σιγά σιγά χάνουμε και την υπομονή μας και τώρα πια πρέπει να βρεθεί μια λύση στο θέμα του ονόματο Τώρα αν θα το πούνε. Άνω Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, η Κάτω Μακεδονία, δεν μπορεί το μέλλον μια χώρα ολόκληρη να εξαρτάται από το όνομα. Όλοι μα και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι πάντα τη λέξη Μακεδονία χρησιμοποιούμε και ω εκ τούτου νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω. Ίσως πλέον ήρθε η ώρα να κερδίσουμε το χρόνο και να σταματήσουμε να καθυστερούμε στην υπόθεση αυτή. Θα παρακαλέσω τώρα τον εισηγητή να λάβει το λόγο για να κάνει κάποιες ακόμα παρατηρήσεις. Μερικές φορές νιώθω υπερήφανος να είμαι μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήθελα να ζητήσω το λόγο. Όχι, επρόκειτο για μια ερώτηση προς τον κύριο Χουντή, αλλά μην ξεκινήσετε τώρα μια συζήτηση ελληνο-ελληνική. Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις οι οποίες απευθύνθηκαν άμεσα σε μένα, λέει ο κύριος Κουμουτσάκος. Για τους Γερμανούς συναδέλφους θα ήθελα να επαναλάβω κάτι το οποίο επανειλημμένα έχω πει εδώ τον στρατηγικό στόχο της Ελλάδας, ο οποίος είναι όλοι οι γείτονές της να ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσετε όλοι. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση, γιατί δεν θα είναι καλό για μας, να υπάρχει μια μαύρη τρύπα στα Βαλκάνια, στον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανένα και ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως προβλήματα υπάρχουν. για τα θέματα που έθεσε η κυρία Ντόρις Πακ, πώς θα τους ονομάζουμε τους ανθρώπους αυτούς. Άκουσε ίσως αυτό που είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Αν θέλει μια απάντηση, να της δώσουν μια απάντηση. Σλάβο Μακεδόνες. Αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα δεκτό. Ιστορικά είναι σαφές, τεκμηριωμένο και σωστό. Τώρα, θα έπρεπε να είχατε την ίδια αντίδραση και όταν πήρε το λόγο το Συμβούλιο. Τώρα για αυτήν την ευαισθησία ε, για μια χώρα η οποία περιμένει 10 χρόνια για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Κοιτάξτε, ορισμένες χώρες πρέπει να έχουν την ίδια ευαισθησία για την Τουρκία η οποία περιμένει 40 χρόνια. Και ξέρουμε ότι οι αντιρρήσεις δεν προέρχονται από χώρες σαν την Ελλάδα αλλά από μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα σε σχέση με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορία. Σχετικά χρειάζεται μια ομοφωνία για να υπάρξει η ιδιότητα, για να αποδοθεί η ιδιότητα ε, του υποψηφίου κράτους. Και η Ελλάδα το έκανε αυτό ελπίζοντας εκείνη την εποχή ότι αυτή η, κίνηση καλής θέλησης θα αλλάξει εν μέρη τουλάχιστον τη στάση των γειτόνων μας οι οποίοι θα έπρεπε να είναι πιο παραγωγικοί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ μας. Αντίθετα, από πλευράς τους τα πράγματα σκλήριναν. Συνεπώς λοιπόν, στην ερώτηση γιατί να αλλάζουμε συνεχώς τη θέση μας, παίρνετε την απάντηση. Τέλος, ο χαρακτήρας του θέματος. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει ένα ψήφισμα του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, πώς το ονομάζεται το θέμα αυτό, διεθνές ή διμερές. Υπάρχει μία σειρά αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Από ό,τι γνωρίζω εγώ την διεθνή σκηνή, έχουμε κατεξοχήν μπροστά μας ένα διεθνές θέμα και ένα τελευταίο θέμα. Γιατί η Ελλάδα, η Αλβανία και η Βουλγαρία είναι ανόητες και πραγματικά ο μόνος σοφός ο κύριος Γκρόσκι. Ναι, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι διαπραγματεύσει με την Τουρκία έχουν ξεκινήσει το 2005, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Χάουιτ έχει το λόγο. Ναι, κρίμα που η συζήτηση σταματάει τώρα. Δεν θα αλλάξω αυτά που ήθελα να πω. Δεν θα ξαναξεκινήσω τη συζήτηση για το ελληνικό θέμα. Το είπα γιατί τέθηκε προφορικό ερώτημα στον συνάδελφό σας. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Χάουιτ. Και ακριβώς είναι και η ένστασή μου. Όταν η κυρία Πακ αναζητά Έλληνες μέσα σε αυτή την αίθουσα και βλέπει μόνο τον κύριο Κουμουτσάκο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχω τίποτα με τον συνάδελφο, You have χρειάζεται μια απάντηση. Σας παρακαλώ, αυτό είναι 15 λεπτά μιλήσατε και δεν σας ε, διάκοψα στην πρώτη σας παρέμβαση. Κύριε Πρόεδρε, προέκυψε στο θέμα. Το λέγω έχει κύριος Χάουιτ. Υπάρχει κάποιος Έλληνας, κάποιος να, να πει είμαι κι εγώ εδώ, είπα κάτι και αν δεν το κατάλαβε κυρία Πακ, θα το επαναλάβω. Ο κύριος Χάουιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κρίμα που σταμάτησε έτσι η συζήτηση. Το συζητάμε μια μισή ώρα τώρα το θέμα αυτό και όπως ε, σας είπα κάποιες μέρες είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή είναι μια τέτοια μέρα γιατί όλοι όσοι παρακολούθησαν τη συζήτηση διαπιστώνουν ότι στη μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού φάσματος στην Επιτροπή μας υπάρχει μεγάλη συμφωνία, μεγάλη συνένεση, μεγάλη συμφωνία. Νομίζω ότι αυτό καταδείχθη σαφώς. Ε, να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους που μίλησαν στο πνεύμα αυτό. Ξέρουμε κύριε Κυρίλοφ, έχετε ε, πολύ ε, έντονες απόψεις, αλλά συνδράματα και συμβάλλατε στη συζήτηση με πολύ ισορροπημένο τρόπο. Κύριε Κουκάν, είσαστε εξαιρετικό ε, εταίρος για τη χώρα αυτή και συμφωνώ με κάθε λέξη που είπατε. Σας ευχαριστώ για τις πολύ στενές αυτές σχέσεις που έχετε μαζί μας και με όλους τους κοιόδης ε, εισηγητής και με τον κύριο Κάτσιν που αναγκαστικά έφυγε και με την κυρία που μίλησα σήμερα. Ελπίζω ότι η ομοφωνία μας να ενισχύσει τα επιχειρήματά μας και αυτό να αποστείλει ένα μήνυμα στα κόμματα της χώρας και στον λαό της χώρας για το πού στεκόμαστε, πού βρισκόμαστε ως χώρα, ως κοινοβούλιο. Πρόεδρε Μπροκ, διάβασα προσεκτικά τα σχόλιά σας και Ακούω την απογοήτευσή σας, όπως την εκφράσατε και στην Ολομέλεια. Σας άκουσα ψεκτικά και στην ε, Ολομέλεια πέρσι και νομίζω ότι η απογοήτευση που εκφράζετε με βρίσκει σύμφωνο. Χαίρομαι που την εκφράζετε ως πρόεδρος της Επιτροπής και νομίζω ότι και αυτό από μόνο το αποτελεί ένα μήνυμα. Να σας πω ότι δεν πιστεύω ότι η εποχή αυτή είναι ε, εθνοτικό ζήτημα πρόκειται ουσιαστικά για διαφωνία μεταξύ των δύο μακεδονικών κομμάτων. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι σοβαρή η διαφωνία αυτή. Να σας ευχαριστήσω για την προσωπική προσοχή που αφιερώσατε, γιατί νομίζω ότι αυτό με βοηθά ως εισηγητή και βοηθά και το Κοινοβούλιο. Όπως είπατε και εσείς και η ε, θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στο θέμα αυτό. Συμφωνώ απόλυτα και προτείνω αναβολή και με τον τρόπο αυτό να αυτό να ακολουθήσουμε. Κανείς δεν θέλει αναβολή, κανείς δεν θέλει να αγοράσουμε επιπλέον χρόνο. Προσπαθούμε να ενεργοποιηθούμε, να ασκήσουμε πίεση για να σημειωθεί πρόοδος. Αυτό που λέω σε εσά Πρόεδρε και σε όλους τους συναδέλφους είναι ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση και σε όλα τα κρατημέλη προκειμένου στο Συμβούλιο να επιδείξουν πολιτική βούληση και ελπίζω ότι και οι χώρες σας και άλλες χώρες να ακούσουν το μήνυμα αυτό γιατί νομίζω ότι και εμείς έχουμε κάνει υποσχέσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τις στηρίσουμε. Ελπίζω το Συμβούλιο να μας ακούσει με πιο πολύ προσοχή, να ακούσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το μέλλον. Τώρα, σε κάποια μεμονωμένα στοιχεία που αναφέρεται κύριε Τάνοκ, βοηθήστε με μήπως ε, δεν είμαι σαφές σε ό,τι αφορά τον, τις τροπολογίες του κυρίου Στογιανόφ. Θα ήθελα να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί το τι εννοούσα αυτά που είπε και αυτός και ο κύριος Πόσελτ το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Κουκάν. Σε ό,τι αφορά την απόφαση αναβολής, δεν θέλουμε η απόφαση αυτή να τύχει λανθασμένης ερμηνείας. Και ο κύριος Κούκαν το ανέφερε. Κάποια κοινή δήλωση της Επιτροπής που θα προσυπογραφεί από τους ε, σκιώδεις. Συμφωνώ να καλέσω τους εκπροσώπους ε, της των, πολιτικών ομάδας, των πολιτικών ομάδων μέχρι αύριο στις 4 να καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία προκειμένου να αποφύγουμε οποιαδήποτε απόπειρα παρερμηνίας των ε, σκοπών μας. Και αυτό δεν θα πρέπει να είναι μονομερές. Εγώ λοιπόν ε, επέλεξα να τοποθετηθώ κατά της αποχής, ξέροντας ότι θα είναι λάθος να κατηγορήσουμε στην, για την κρίση αυτή μόνο ένα κόμμα. Ελπίζω να γίνει κατανοητό ότι η ευθύνη για την κρίση αυτή βαραίνει όλα τα κόμματα. Δεν εννοούμε ότι δεν είναι όλα τα κόμματα υπεύθυνα. Για τον κύριο Κουμουτσάκο και για κάποιους άλλους. Αυτό που λέω μόνο είναι ότι κάποιες φορές στο κοινοβούλιο αυτό δεν ακούω παρεμβάσεις που ακούω όταν είμαι στην χώρα και σε γειτονικέ χώρες. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο να επιληθεί το θέμα του ονόματος, αλλά έχουν σημειωθεί τεράστιες πρόοδοι, κοιτώντα τις ανταλλαγέ που έχουν λάβει χώρα και με τον ε, Βούλγαρο Υπουργό Εξωτερικών στα Σκόπια. Πράγματα που δεν θα μπορούσαν να έχουν συμβεί πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει αυτό να το ενθαρρύνουμε, όχι να το αποθαρρύνουμε. Και αυτό το λέω και προς τους συναδέλφους στην Επιτροπή. Ευχαριστώ τον κύριο Μπράνκοβιτς για την ε, παρέμβασή του. Πολύ σωστή και στέλνει ένα πολύ καλό μήνυμα προς όλους. Τον ευχαριστώ. Νομίζω ότι δίκαιο είναι να τονίσουμε ότι όντω τα πρακτικά ότι ο διάλογο πολιτικού υψηλού πολιτικού επίπεδου δεν αντικαθιστά τι διαπραγματευτικέ διαδικασίε. Πρόκειται για ένα κλειδί που θα ξεκλειδώσει ίσω τι ε, συνομιλίε για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Προ την κυρία Μπρισάτζιτ. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα να προφέρω το όνομά σας καλύτερα. στην προφορά τα πηγαίνω καλύτερα από τον Πρόεδρο. Αλλά έχετε δίκιο. Η ανάλυση σας είναι εξαιρετική και θα πρέπει να την ακούσετε. Πολεμούμε στην περιοχή αυτή με αντίπαλο τον εθνικισμό. Και στις χώρες για τις οποίες κάνω εκθέσεις, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος του εθνικισμού. Έχετε δίκιο για την ανησυχία σας αυτής που εκφράζεται. Σας ευχαριστώ που τα αναφέρετε αυτά. Και πρόεδρε, κλείνοντας να πω το εξή. Και αυτό το είπα πριν από καμιά εβδομάδα στην ίδια τη χώρα. Ελπίζω αυτή η συζήτηση να αποστείλει ένα θετικό μήνυμα ότι είμαστε υπέρ του ευρωπαϊκού μέλλοντος και της ευρωπαϊκής μοίρα της ε, χώρας, αλλά δεν δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της χώρας αν ο ίδιος ο λαός, η ίδια, τα, τα ίδια πολιτικά κόμματα δεν το θέλουν ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η πρόκληση. Αυτή είναι η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα και στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθούν. Σας ευχαριστώ. Έχουμε νομίζω συμφωνία να αναβληθεί η ψηφοφορία για μία μόνο σύνοδο. Γιατί δεν θα πρέπει να ε, δώσουμε ευκαιρίες σε αυτούς που απέχουν και θέλουν να παραποδίσουν εργασίες του Κοινοβουλίου ε, με μια έκθεση που αφορά το 2011. Αναβάλουμε λοιπόν και κυρίως το πέρασε των εργασιών της Επιτροπής μας. Το, ε, κυρίσω μάλλον ε, το τέλος του θέματος αυτού και κάποιο συνάδελφος ζήτησε τον λόγο για μια προσωπική δήλωση, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, εκ του γεγονότος ότι στην προηγούμενη διαδικασία δεν μου δόθασε την ευκαιρία να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα, στην συμφωνία περί να αναβληθεί η, ψήφιση της έκθεσης να αποσύρετε την συμφωνία της ΓΚΟΕ. Έχετε, έχετε το λόγο για... Αναβολή της ψήφισης. Ja, dann, dann äh, hat... Άρα η ομάδα της ΓΟΕ δεν υποστηρίζει την απόφαση αυτή. Και πάμε στο σημείο 7. Δικαιώματα των γυναικών στις υποψήφιες βρετανικές χώρες. Με την κυρία Μποσκούρτ, ως συντάκτρια γνωμοδότησης, η κυρία Γκόμες. Η κυρία Μποσκούρτη είναι η συγγήτρια, δεν μπορεί να είναι μαζί μας όμως σήμερα. Μου άφησε τις σημειώσεις της, τις οποίες θα σας τις διαβάσω. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα κεντρικό θέμα για τις διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Και δεν θα πρέπει να αντίθεται απλά σε μία ή δύο παραγράφους με σύντομες αναφορές. Θα πρέπει λοιπόν να είναι προτεραιότητα στις εκθέσεις μας για τις χώρες αυτές. Οι χρηματοδοτήσεις προς τις χώρες αυτές θα πρέπει να στοχεύουν και στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή και να ενθαρρύνεται το επιχειρηματικό πνεύμα των γυναικών. θα πρέπει να καταπολεμάται η οικιακή βία, η υποχρεωτική πορνεία ε, και η παιδική εργασία είναι απαράδεκτες καταστάσεις που πρέπει να καταγγελθούν. Θα πρέπει να υπάρξουν προσπάθειες για την αποκατάσταση των θυμάτων της βίας ατομικής ή ομαδικής στις περιοχές αυτές. Ε, η συγγήτρια ε, μπορεί να χαιρετήσει ε, τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε κάποιες τουλάχιστον από αυτές σε συμβιβαστική λύσεις, τις οποίες θα προτείνουμε μέσω των τροπολογιών μας για θέματα σώματεμπορίας, σαν παράδειγμα, για θέματα καταπολέμησης οικιακής βίας κτλ. Σε ευχαριστώ. Υποστηρίζω την κυρία Γκόμες ασφαλώς. Η έκθεση είναι πολύ καλή. Οι τροπολογίες συχνά είναι διπλές και τριπλές και γι' αυτό θα πρότεινα η συγκήτρια να ψάξει συμβιβασμούς στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών. Θα πρέπει να τύφεται και το θέμα των δικαιωμάτων της γυναίκας και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και θα έπρεπε να παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ότι ως τώρα. Είμαι κάπως διστακτική σε ό,τι αφορά ότι θα πρέπει να αποτελεί αυτό προτεραιότητα στην έκθεση πρόοδου. Ίσως αυτό να είναι λίγο παρατραβηγμένο, αλλά θα πρέπει να παίζει ένα ρόλο, σύμφωνοι. Να τονίσουμε επίσης σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των γυναικών ε, στην ε, κοινωνία των πολιτών, και στι πολιτικές δραστηριότητε θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και στις δυτικέ μας χώρες. Θα πρέπει να το ε, θίξουμε εξ αρχής. Και χαίρομαι που στο σημείο 9 μιλάτε για την αποκατάσταση των θυμάτων στα Βαλκάνια. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Βοσνία-Ζεγοβίνη. θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει οι επιτόπου φορείς και παράγοντες να επιβάλλουν τη δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτό είναι ανοησία. Έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά σε ό,τι αφορά την έβρεση θέσης εργασίας. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευρά δική μου θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Νομίζω ότι γενικά υπάρχει ευρία σύμφωνία για τα θέματα που ανέφερε και η Αναγκόμε και η Doris Πακ. Να αναφέρω ωστόσο κάποιες τροπολογίε που καταθέσαμε και νομίζω ότι και άλλες ομάδες ε, κατέθεσαν τροπολογίε, σημαντικέ ε, τροπολογίε σε ό,τι αφορά τι γυναίκε θύματα εγκλημάτων πολέμου βιασμών κλπ. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της έκθεσης. Επίσης ε, κατέθεσα μια τροπολογία για την εφαρμογή των ποσοστώσεων. Έχουμε κάποια καλά παραδείγματα στο Κωσυφοπέδιο και στο Μαυροβούνιο όπου έχει σημειωθεί πρόοδος για να βελτιωθεί η εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα τα πολιτικά. Μια τροπολογία επίσης για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων σε ό,τι αφορά και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, πολέμηση της ομοφιλοφοβίας σε όλες τις ε, περιοχές αυτές. Νομίζω ότι εν γέννη είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η συμβολή της Επιτροπής ε, της δικής μας. Δεν νομίζω όμως να υπάρχουν ουσιαστικά ιδιαίτερες διαφωνίες με την ε, καθήλια αρμόδια Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι καλή η έκθεση και θα βρούμε και καλές συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Χουντής. Ε, ελπίζω να μας ε, βοηθήσετε όταν συμφωνεί η κυρία Λούνατσα και η κυρία Γκόμες και η κυρία Πάκ. Ε, εγώ έχω λίγο νευρικός, δεν έχω κοιτάξει την έκθεση. Ίσως θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε και να διευκρινίσετε την κατάσταση. Να υπάρχει ελπίδα και για τα Βαλκάνια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην πρόθεσή μου να βοηθήσω Απλώς προλίγου η αψημαχία μας ήταν ότι και εσείς δεν βοηθούσατε, σε ποιο πράγμα δεν βοηθούσατε και θα δείτε ότι εδώ όταν γίνεται μια συζήτηση δεν συζητάνε μόνο οι μεγάλες ομάδες. Συζητάνε και οι μικρότερες, τουλάχιστον με τα σημερινά αποτελέσματα ομάδες. Ένα. Και πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και αυτό το στοιχείο. Δεν έχω καμία πρόθεση να επαναφέρω αυτό το θέμα. Πάω στην ουσία της έκθεσης για να πω ότι η Γκουε, η ομάδα μου, ως σκιώδης συγητής που είμαι, συμφωνούμε με την έκθεση της συναδέλφου, πιστεύουμε πως είναι σε θετική κατεύθυνση και ότι το πρόβλημα αυτό είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό και για τις Βαλκανικές χώρες που είναι υπό ένταξη. Δύο-τρεις σύντομες παρατηρήσεις, πάλι στο πνεύμα να βοηθήσω την ε, υπόθεση και όχι να το δυσκολεύσω. Το πρώτο που έχουμε παρατηρήσει και που εκεί πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση είναι ότι σε αρκετές από αυτές τις χώρες που είναι σε ε, ενταξιακή διαδικασία, ενώ λαμβάνονται κάποια σωστά μέτρα, ενώ ψηφίζονται ορισμένοι σωστοί νόμοι όσο αφορά τη θέση της γυναίκας, δεν εφαρμόζονται. Και το πρόβλημα λοιπόν της εφαρμογής αυτών των σωστών μέτρων είναι πάρα πολύ σημαντικό, το συναντάμε σε όλες τις, ε, τις χώρες. Και επομένως, στη διαδικασία ένταξης η απέτηση το θέμα των ε, ε, γυναικών της αναβάθμισής του, της ίσης ε, μεταχείρισης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η δεύτερη μου παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, και θα τελειώσω, διότι υπάρχουν, βλέπω και άλλα θέματα, είναι πως για να λυθούν μια σειρά θέματα, τα οποία εντοπίζει η συνάδελφο η συγγήτρια, αλλά και το ψήφισμα της κυρίας Κορνέλιασεν, πρέπει να λυθούν σε βάθος χρόνου κάποια πιο, θα έλεγε κανείς, βαθιά διαχρονικά ζητήματα. Αναφέρομαι ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό τι θέλω να πω και τελειώνω. Έχουμε το πρόβλημα της ε, ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, το θέμα της πορνείας, που είναι μια μορφή όμως έκφρασης του οργανωμένου εγκλήματος, που δυστυχώς έχει πάρει μεγάλη έκταση στα, στην περιοχή των Βαλκάνιων και ενδεχομένω και άλλο. Άρα στις ενταξιακές εκθέσεις που θέτουμε τέτοιο θέμα να ξέρουμε ότι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος θα έχει θετικές παρενέργειες και σε μια σειρά σημεία που εντοπίζει η έκθεση τη συναδέλφου. Τελείωσα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστώ κύριε Χουντή. Το κατάλαβα ότι δεν θα με βοηθούσατε στο θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δικαίωμά σα για το πρώτο θέμα. Λάβατε το λόγο πριν από ομάδες που είναι μεγαλύτερες από ε, εσάς και μιλήσατε πολλή ώρα για το θέμα ε, αυτό, όπως και ο εισηγητής σχεδόν τόσο πολύ. Σας παρακαλώ λοιπόν την κατανόησή σας για το ότι δεν ξαναπήρετε το λόγο. Και περνάμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε το θέμα αυτό. Στις 4 Μαρτίου ψηφίζεται στην Επιτροπή μας το θέμα αυτό. γιατί στην Ολομέλεια προβλέπεται για τον Απρίλιο. Περνάμε τώρα στο 8, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Ο τσαν στανοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. μετά την ανακοίνωση που κάνατε για τον κύριο Κασουλίδη, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, πέντε υπουργοί των 27 χωρών είναι τέως ευρωβουλευτές. Κάτι σημαίνει αυτό. Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο και ε, Κύπρος. Και φυσικά έχουμε τρεις πρωθυπουργούς μεταξύ μας είναι και ο κύριος Κουκάν. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε άλλες τέτοιες ενδιαφέρουσες στατιστικές Πέρα λοιπόν από την τεχνική θα έλεγα διαδικασία που έχετε μπροστά σας, είδα πώς γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι εμπορικές ποσοστώσεις και ε, προσπάθησα να καταλάβω γρήγορα και είδα ότι η λαϊκή Κίνα έχει δικαίωμα μια αντισταθμιστική ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με τις απώλειες που σημειώθηκαν εις βάρος της ε, ε, λόγω της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Τελωνιακή Ένωση. Θεωρητικά λοιπόν η Κίνα χάνει εν μέρη ε, την πρόσβασή της σε αυτές τις αγορές και γίνεται μια πρόταση ρυθμίσεων η οποία θεωρείται μια έλογη μορφή αντιστάθμισης ε, της ε, απώλειας ε, της λαϊκής δημοκρατίας. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι δεν έχω καμία, μετά από εξέταση του θέματος, δεν έχω καμία επιφύληξη για να υποστηρίξω την πρόταση της Επιτροπής μας για να ζητήσει από την αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου και από το σύνολο του Κοινοβουλίου να συμφωνήσουν με την συγκεκριμένη πρόταση σε επίπεδο συνθήκης της Λισαβόνας υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή και να επικυρωθεί τάχιστα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σύντομος και συνοπτικός. Ο υπολογισμός αυτός ε, τρεις ε, πρώην ε, πρόεδροι είναι, του Κοινοβουλίου είναι μέλη της Επιτροπής μας. Μπούσεκ, και Να δούμε πόσοι υπουργοί εξωτερικών, πόσοι πρωθυπουργοί, πόσοι επίτροποι ήταν μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Να σας πω μια ιστορία πριν από κάποια χρόνια. Ο πρόεδρος ε, υπουργός, ο πρόεδρος πρόεδρος, ο γερμανός πρόεδρος είπε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει ε, θέματα εξωτερικής ασφάλειας. Και είπα ότι συμφωνώ. ότι κανείς ε, πρόεδρος της Επιτροπής δεν μπορούσε να το κάνει αυτό εκτός από τους ε, πρώην πρόεδρους εξωτερικών και τους πρωθυπουργούς. Είναι ένα θέμα το οποίο συχνά δεν είναι γνωστό στο κοινό και νομίζω ότι θα πρέπει να το προβάλλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τσάρλς, για την υπόδειξη αυτή και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κουκάν. Κύριε Κουκάν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρου του κυρίου Γκουριάνου και συζητητού του Ευρωπαϊκού Λεκόμματο που δεν μπορούν να είναι παρόν εδώ, μεταφέρω το μήνυμά του, απλό, θετικό, σύντομο. Ευχαριστούμε τον κύριο Τάνοκ για την γνωμοδότηση. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει την πρόταση της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας με την προσαρμογή των δαγμολογικών δασμών μετά την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θεωρεί ότι πρόκειται για ένα αγκαίο τεχνικού χαρακτήρα βήμα για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και για την ε, διαμόρφωση απρόσκοπτων σχέσεων με την λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Ταυτόχρονα καταγράφει τη σημασία και των θημερών εμπορικών ε, κανόνων και υπογραμμίζει την ε, προσήλωσή της στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου εισηγητής λοιπόν έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο πιστεύει ότι μπορεί να προχωρήσει για υποβολή στην αρμόδια καθήλη επιτροπή η γνωμοδότηση αυτή. Σα ευχαριστώ πολύ. Τρεις ακόμη πρωθυπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί. Ο κύριος Φερχόφστατ, ο κύριος Δεχάνε. Και ένα τρίτο που δεν ε, μπόρεσαν οι διερμηνεί σα να αναγνωρίσουν είναι επίση μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ θερμά. Έχουμε τίποτα στα διάφορα. Όχι, σα ευχαριστώ και χαίρετε. Καλό σα βράδυ. Με κάθε ευτυχία. Και από ό,τι φαίνεται, ο Πέπε Γκρίλο και ο Μπαρλουσκόνη θα έχουν την πλειοψηφία στην Βουλή στην Ιταλία. Στη Γερουσία στην Ιταλία. Δεν είναι πολύ σαφή η εικόνα ακόμη, αλλά προ το εκεί τίνει.